Mes chers collègues, j'ouvre. Euh, Συνάδελφοι, καλημέρα. Ξεκινάμε. Έχουμε μια πολύ πυκνή ημέρα μπροστά μας και πλούσια μέρα. Θα έχουμε την τιμή να υποδεχθούμε τον Επίτροπο Έτιγκερ ο οποίος ε, είπε ότι θα είναι παρόν σήμερα όταν συζητήσουμε τις βασικές γραμμές των συναδέλφων Τομά και για το πολιετές δημοσιονομικό και την έκθεση Λεβαντόσκη και Ντεπρέ για τους ίδιους πόρους. Δύο θέματα τα οποία συνδέονται φυσικά μεταξύ τους και εμείς πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρξουν νέοι πόροι δεν μπορεί να υπάρξει νέο πολιετές δημοσιονομικό. Είναι η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς πάντως και θα ήθελα να σας μεταφέρω τις καλύτερες ευχές μου και προς εσάς κύριε Επίτροπε και για τη δράση την οποία αναλαμβάνετε και για την οικογένειά σας και για όλους εσάς, τους συνεργάτες, τους συμβούλους, τη γραμματεία Ελπίζω η φετινή χρονιά να είναι μια ενδιαφέρουσα, ευτυχισμένη χρονιά. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Το πολιετές δημοσιονομικό για την περίοδο μετά το 20, οι τελευταίες διαπραγματεύσεις για το Brexit, οι ήδη οι πόροι, μια ολόκληρη σειρά προκλήσεων και το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους και για όλους. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ τον Γενικό Εισηγητή που δέχτηκε να αναβάλουμε τη συζήτηση για την έκθεσή του για να επωφεληθούμε από την παρουσία του κυρίου Έτιγκερ για τα θέματα των ιδίων πόρων. Η ημερήσια διάταξη γίνεται συνεπώς δεκτή. Να σας υπενθυμίσω ότι οι αποφάσεις των συντονιστών της 4ης και 11ης Δεκεμβρίου του 2017 βρίσκονται στο φάκελό σας και αν δεν έχετε αντιρρήσεις θεωρώ ότι όσοι είναι διατυπωμένες αυτές οι αποφάσεις θεωρούνται αποδεκτές. Να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 6.30 σε αυτή την αίθουσα θα προσφερθεί ένα κοκτέιλ για την αρχή του χρόνου και όπως έχουμε βάλει τις ψηφοφορίες λίγο πριν το κοκτέιλ σημαίνει ότι θα είναι πολλοί παρόντες. Θα ήθελα επίσης να είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά της συνεδρίας της 4ης Δεκεμβρίου. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται δεκτά. Περνάμε στο 5 και 6 τα οποία θα αντιμετωπίσουμε από κοινού την παρουσία του Επιτρόπου. Θέλω για μια ακόμη φορά να τον ευχαριστήσω εξ ονόματός σας για την παρουσία του. Είχε προβλέψει να είναι απόν και από την συνεδρίαση των Επιτρόπων αλλά η μερίσια διάταξη δυστυχώς τον υποχρεώνει να είναι εκεί και θα πρέπει να φύγει στις 10.30. Όταν οι συνεισηγητές μας για το πολιετές δημοσιονομικό και για τους ιδίους πόρους ε, μιλήσουν, θα μιλήσει και ο Επίτροπος. Θα γίνει μια συζήτηση με το σύνολο των μελών με τους σκιώδεις, με τους γνωμοδότες και τέλος με τους συντονίστες και τα υπόλοιπα μέλη. Όπως σας είπα στις 10.30 θα φύγει ο Επίτροπος. Και φυσικά Επίτροπε θα έχετε το λόγο όποτε το επιθυμείτε έτσι ώστε η συζήτηση να είναι πράγματι ενδιαφέρουσα. Δίνω λοιπόν για πέντε λεπτά το λόγο στο, στους συνεισηγητές. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Όλμπριχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εφόσον συμφωνεί και η κυρία Τομά, θα κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα περάσουμε στην κυρία Τομά για το δεύτερο τμήμα. Η έκθεσή μας είναι το επόμενο βήμα, αν θέλετε, για το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το θέμα δεν είναι μόνο το πολιετές δημοσιονομικό, αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο. Εμείς στην ουσία για μια ακόμη φορά αντιδρούμε στην θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατετέθη στα πλαίσια της Δευκής Βίβλου για το μέλλον των δημοσιονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κρέτσου. Και υπήρχαν ορισμένα ερωτήματα στην ανακοίνωση αυτή για κάποια πιθανά σενάρια, εξελίξεις, θεμένη αξία κτλ. Πήραμε λοιπόν το έγγραφο αυτό πάρα πολύ σοβαρά και δεν θέλουμε μόνο να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό, αλλά να θέσουμε θέματα όχι μόνο στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και την θέση μας την τελική πριν την άποψη της Επιτροπής τον Μάιο. Να ενημερώσουμε το Συμβούλιο τι μπορεί να περιμένουν από μας όταν μας προτείνουν τις θέσεις τους τελικά Οι θέσεις μας λοιπόν δείχνει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα παρετηθεί από τις φιλοδοξίες, όχι τις φιλοδοξίες του Κοινοβουλίου, αλλά τις φιλοδοξίες της Ένωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι έχει φτάσει η στιγμή, ιδιαίτερα μετά το Brexit, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι πριν από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να διατηρήσουμε τις πολιτικές τις οποίες έχουμε. Φυσικά και είμαστε υπέρ της απλοποίησης, φυσικά και είμαστε υπέρ διορθωτικών κινήσεων, αλλά οι πολιτικές αυτές λειτουργούν. Ιδιαίτερα πολιτικές ε, όπως η περιφερειακή, η γεωργία, υπάρχουν θέματα στην εφαρμογή τους. Θα πρέπει όμως να διατηρήσουμε τις πολιτικές αυτές και συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν και νέες προτεραιότητες και νέες προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στου στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, στο μελλοντικό ε, πολιετές δημοσιονομικό, δηλαδή μετανάστευση, άμυνα, η μετανάστευση έχει δύο διαστάσεις. Μία εσωτερική διάσταση, τι θα κάνουμε με τους μετανάστες τους παράτυπους και δεύτερον τι θα κάνουμε έτσι ώστε στο μέλλον να αποφύγουμε τη μαζική αυτή μετανάστευση η οποία μπορεί να είναι εκτός ελέγχου. Εφόσον έχουμε προτεραιότητες λοιπόν και εφόσον συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρούμε τους επιπλέον πόρους. Επιπλέον πόρους είναι νέες προτεραιότητες εμείς σαν εισηγητές δεν προτείνουμε οι παλιές πολιτικές να αντικατασταθούν από τις νέες. Εμείς πιστεύουμε ότι οι νέες προοπτικές απαιτούν νέους πόρους. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα συμβατό με αυτά τα οποία έχει παρουσιάσει ο κύριος Σέτιγκερ. Για την αρχή της συζήτησης εμείς πιστεύουμε, θεωρούμε ότι η συνοχή, η περιφερειακή πολιτική και η ε, γεωργική πολιτική θα πρέπει να παραμείνουν στο σημερινό ονομαστικά επίπεδο. Με την μείωση φυσικά της, Ευρωπα... Ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Προτείνουμε λοιπόν το Horizon 2020 το Erasmus Plus ε, και το Doubling ε, να αυξηθούν σε ποσοστό. New priorities. As a consequence, as a consequence, according to our very, very general analysis. Ε, να διπλασιαστούν λοιπόν κάποια ταμεία και αυτό κάνει εντύπωση, αλλά είναι καρπός μιας πολύ σοβαρής ανάλυσης. Εμείς πιστεύουμε ότι το πολιετές ε, δημοσιονομικό θα πρέπει να βασίζεται στα, στο ακαθάριστο ε, ποσοστό 1,3. Ε, δεν είναι μη ρεαλιστικό αυτό. Σαν παράδειγμα συζητάμε για 1,2 δίσκα τέτος για την άμυνα. Αυτό καταλήγει στο 1,3% του κοινοτικού ΑΕΠ. Ξέρω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 1,1 συν. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο 1,2. Εμείς προτείνουμε σαν κοινοβούλιο ε, να προτείνουμε το 1,3. Ξέρω ότι υπάρχουν ανάγκες ε, για τις αλλαγές της πολιτικές, για τις διαφορετικές πολιτικές, για να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι πολιτικές. Αλλά θα πρέπει να δούμε επίσης και ποιες είναι οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Ευχαριστώ η κυρία Τωμά. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω κύριε Επίτροπε. Θα αναφερθώ σε πιο τεχνικές πτυχές σχετικά με τις ε, δικές μας απαιτήσεις για την ε, δόμηση του προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος ε, το έχει πει επανειλημμένος ότι υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες θα πρέπει να τύχουν σεβασμού ε, καταρχήν η ενότητα Τα εξωτερικά ταμεία θα πρέπει να ενταχθούν στον προπολογισμό. Η... Ο ισοσκελισμός του προπολογισμού και ο ισοσκελισμός ανάμεσα στις ε, πληρωμές και τα έσοδα. Ε, η καθολικότητα, δηλαδή ε, όχι δικιά έσοδα για συγκεκριμένες δαπάνες. Και τέλος, η, ε, ο σεβασμός του άρθρου 311, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για να καλύψει τις πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες έχει καθορίσει. ένα άρθρο το οποίο το έχουμε ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό. Μετά ε, θα θέλουμε να δούμε το θέμα της διάρκειας και της συμβατότητας ε, το, της θητείας του Κοινοβουλίου με την θητεία της Κομισιόν καθώς και σε σχέση με τη διάρκεια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχει διάρκεια 7 ετών αλλά θα θέλαμε στο κείμενο να αναφέρεται ότι από την επόμενη θητεία ε, θα πρέπει να γίνεται μια ενδιάμεση αναθεώρηση ε, στα πέντε χρόνια με ένα πολιετές δημοσιογραφικό πλαίσιο που θα διαρκεί δέκα χρόνια. Έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ε, ε μακροπνοού σχεδιασμού. Θυμάστε αυτή τη συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ και αρκετό, κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Συνεπώς ενδιάμεση αναθεώρηση το μέσον της διάρκεια. αύξηση τη ευελιξίας, την έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα, αλλά θέλουμε να την ενισχύσουμε. Το κάναμε στην αναθεώρηση του 2016, με μια χρησιμοποίηση ε, πόρων ε, σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση. Καθώς επίσης ε, και όταν συζητούσαμε, ε, συγγνώμη, ζητάμε επίσης αύξηση του προπολογισμού των, ε, στα 2 δισεκατομμύρια για την ευελιξία, καθώς επίσης και αύξηση των ποσών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελεγγύης. έχουμε λάβει υπόψη τις προτάσεις σας για το θέμα της προσθέμενης αξίας συμφωνούμε και θα πούμε στο κείμενο ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη διευκρίνηση. Γιατί το στη συζήτηση της Επιτροπής μας ε, έγινε σαφές ότι η προσθέμενη αξία μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και εμείς στηρίζουμε και επιθυμούμε απλοποίηση των πολιτικών. Και βέβαια έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα της διαφάνειας. Η σημερινή σας συνάντηση της Κομισιόν για την ε, χρηματοδότηση της ε, Τουρκίας δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε πολύ πρόοδο. Γιατί την... είχαμε πει στις διαπραγματεύσεις ότι το... Ε, δεν είχαμε πει ότι το απόθεμα θα χρησιμοποιείται για την Τουρκία. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια λοιπόν στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται σε σχέση με το, με το Κοινοβούλιο. Για την κρίση των πληρωμών είχαμε πει ότι η, οι πιστώσει πληρωμών θα πρέπει να πλησιάσουν περισσότερο στις ε, πιστώσει ανάληψης υποχρεώσεων. Και ένα άλλο θέμα, το οποίο θα συζητηθεί πολύ εδώ νομίζω, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Η δομή του προϋπολογισμού θα πρέπει να συνάδει με τις πολιτικές προτεραιότητες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, οπότε χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Δεύτερον, συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα και να ενισχυθεί η διάρκεια της. Τρίτον, συνοχή και αλληλεγγύη θα πρέπει να ενισχυθούν στον προϋπολογισμό, να γίνουν κεφάλαιο Τρίτον, το θέμα της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο θα πρέπει να είναι επίσης αντικείμενο κεφάλαιο ξεχωριστού. Η ασφάλεια και η ειρήνη είναι μια καινούρια προτεραιότητα που επίσης μπορεί να γίνει κεφάλαιο. Και βέβαια η διοίκηση αναπόφευκτο κεφάλαιο. Το σημαντικό είναι να μην δημιουργηθεί η πολιτική σύγχυση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν στον ίδιο τομέα να έχουμε την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Γιατί αλλιώς δημιουργείται μια πολιτική σύγχυση που ε, δεν είναι ωφέλιμη. Τόσο στη δημοσιότητα όσο και στη διαχείριση των πόρων. Το θέμα της ε, Τουρκίας, της ε, ε διευκόλυνσης για την Τουρκία. Ε, έχω αιμονή με αυτό αυτό που θα μπει στην μετανάστευση ή στην θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Χρειάζεται λίγο περισσότερη ε, ευκρίνεια σε αυτά τα πράγματα. Τελειώνω, Πρόεδρε. Τελειώσα. <laughs> Ε, η συζήτηση όμως θα συνεχιστεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Τωμά. Όλα αυτά θα κάνουν πιο ειλικρινή και αληθινό τον προπολογισμό. θα περάσουμε στους συνεισηγητές των ιδίων πόρων. Ο κ. Ντεπρέ, πρώτος, ο, και ο κ. Όλμπριχτ θέλει να πει δύο λόγια για τη διαδικασία. Έχουμε ένα κεφάλαιο για τις ε, τομεακές πολιτικές που είναι αποτέλεσμα των, της γνώμης των διαφόρων άλλων επιτροπών Πρόκειται για μια εισαγωγή στη συζήτηση για τους νομιακούς κανονισμούς. Δεν έχει σχέση με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί θα δούμε με τους ηγητές, μπορεί να αλλάξει το κείμενο. Και το σημαντικό για μας είναι η διαδικασία. Πότε θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Αυτό είναι σημαντικό γιατί εμείς θέλουμε να τελειώσουμε πριν τις εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια δυναμική που να μας οδηγήσει να τελειώσουμε πριν τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο στο τέλος. Πρόεδρος, ε, θα δώσω το λόγο στους δύο συνσηγητές για τους ίδιους πόρους. Ε, Ζεράν Ντεπρέ. θα περιοριστώ σε κάποιες ε, γενικές αρχές για τις οποίες υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ ε, του κυρίου Λεβαντόφσκη και μου του ιδίου. Πρώτο σημείο στο οποίο επιμένουμε. Το Κοινοβούλιο χρειάζεται να, έχει, να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο ανάμεσα στην αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και στους νέους ίδιους πόρους. Γιατί όταν δούμε τη διαδικασία για τους ίδιους πόρους, ο, ο, ρόλος του Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά περιορισμένος, παρόλο που είναι πολύ πιο ισχυρός στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική σύνδεση μεταξύ των δύο, δεν θα πετύχουμε και πολλά πράγματα. Δεύτερον, αναλύσαμε με τον κύριο Λεβαντόφσκι την έκθεση της ομάδας ψηλού επίπεδου του, την ομάδα, της ομάδας Μόντι δηλαδή και κάνουμε τις παρατηρήσεις μας με βάση αυτήν. Είναι μια πολύ λεπτομερής μελέτη, ε, πολύ έγκυρη μελέτη και είναι ένα έγγραφο το οποίο αποτελεί αντικείμενο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ των τριών βασικών θεσμικών οργάνων. Τρίτον, προτείνουμε καινούριους ίδιους πόρους με βάση τις εξής αρχές. Θα είναι ένα πακέτο μια δέσμη, έτσι ώστε να είναι ισορροπημένη. Δεύτερον, αυτή η δέσμη θα έχει τρεις στρατηγικούς στόχους που αντιστοιχούν στο ευρωπαϊκό ε, κοινό συμφέρον και έχουν προστιθέμενη αξία. Τρίτον, οι νέοι διπόροι δεν θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν όλοι μαζί, αλλά σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες τι προτεραιότητες και τι πρακτικέ δυνατότητε εφαρμογή. δυνατότητες Τέταρτον, αυτοί οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να ισχύσουν παράλληλα με το σύστημα που ισχύει ως τώρα, με αυτούς τους πόρους ε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που είναι οι τελωνιακοί δασμοί, οι αγροτικέ φορές κλπ. Τέταρτον, ε, ε, θα πρέπει να καταργηθούν οι μειώσει και οι μειώσει των μειώσεων. Παρόλο ότι κάποιοι μηχανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν διορθωτικά. Έκτον, η σφορά, οι κρατικές σφορές θα διατηρηθούν σε κάποιο ποσοστό ε, ως τμήμα του προπολογισμού. Και τέλος, δύο σημαντικές αρχές μας οδήγησαν, μας καθοδήγησαν. Πρώτον, να διατηρηθεί ε, η, η κρατική αρμοδιότητα για το φορολογικό σύστημα και Δεύτερον, οι νέοι ήδη πορεί θα πρέπει να επιβληθούν ε, ε, θα πρέπει να ισχύσουν με παράλληλη μείωση των κρατικών εισφορών από τους προπολογισμού των κρατών μελών. Αυτές είναι οι βασικές αρχές σε οποίες έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο Λεβαντόφσκι. Λεβαντόφσκι. Ο κύριος Λεβαντόφσκι τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με την έκθεση αυτή ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο. Ένα νέο κεφάλαιο σε αυτήν ε, την ατελείωτη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διορθώσει την πλευρά των εσόδων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Και εδώ πέρα έχουμε το παράδοξο των Ευρωπαϊκών Δημοσιονομικών. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο υπόκειται σε μεγάλη κριτική, αλλά το οποίο είναι αρκετά σταθερό. Άρα πρόκειται για μία ακόμα απόπειρα, δεδομένου και του ότι με το Brexit έχουμε μία ευκαιρία να <clears throat> μειώσουμε κάποια από τα ζητήματα που ανακύπτουν. Φυσικά βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο και ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε το τι προτείνουμε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο αυτό θέμα των ίδιων πόρων. Το να είμαστε προσεκτικοί σημαίνει να μην προτείνουμε αλλαγέ συνθήκων, όπως ανέφερε και ο Ζεράρ. Διατηρούμε την δημοσιονομική επικυριαρχία των κρατών μελών. Χρειάζεται ομόφωνη λοιπόν απόφαση και επικύρωση από τις ε, εθνικές βουλές και δεν υπάρχει και ρήτρα πασαρέλ και δεν υπάρχει το θέμα της ε, φορολογίας που συνδέει τους ευρωπαϊκούς πολίτες με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί προσπαθούμε να αποφύγουμε την ορατότητα των ζητημάτων αυτών σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Νομίζω ότι καλό είναι να μην τα κάνουμε αυτά ιδιαίτερα ορατά στους λογαριασμούς των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει ασφαλώς να επιλεγεί, να επιλεχθεί ε, ένα σύνολο νέων ε, προτάσεων. Κάποιε από τι προτάσει αυτέ τι έχουμε ξαναδεί σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, για παράδειγμα. Ο ΦΠΑ φαίνεται να είναι πιο εναρμονισμένο φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 21,5% κατά μέσο όρο. Από 17% στο Λουξεμβούργο μέχρι 27%. Είναι μεγάλο το περιθώριο. Ο βασικός συνελιστής λοιπόν θα έπρεπε να είναι πιο σημαντικός και όχι τόσο πολύ η μείωση που είναι συχνή σε διάφορα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διαγράψουμε πάνω από 12 έως 13% των εσόδων στον προπολογισμό σε σχέση με σήμερα. Η δεύτερη πρόταση, την οποία επίσης την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, το 2011 έγινε η πρόταση αυτή, είναι το FTT. Αυτός ο φόρος των δημοσιονομικών ε, συναλλαγών, όχι ο φόρος δημοσιονομικών, ε, δημοσιονομικής δράσης. Και μην τον παρελέξουμε. Μιλάμε για συναλλαγές, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Γιατί συχνά μιλάμε για τον φόρο Πού προτέθηκε το 1970 ε, με το σύστημα Bretton Woods που κατέρευσε. Αυτό έχει τότε προταθεί ως αντίδραση. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να προτείνουμε αυτό που είχαμε προτείνει και το 2011 για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να μην ε, είναι υπερβολική η επιβάρυνση με φορολόγηση των οικοκυριών. Αν κάποιος δηλαδή δανείζεται για καταναλωτικούς σκοπούς, ε, για στέγαση, να μην είναι υπερβολική η επιβάρυνση φορολογική και να φορολογούνται σωστά και μικρομεσαίες. Και νομίζω ότι ε, έτσι μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός, πέρα από την ε, ενισχυμένη συνεργασία. Επόμενο κεφάλαιο, η εταιρική φορολόγηση, περίπου 1 ή 2% της ε, εταιρικής φορολόγησης. Με τις προσπάθειες εναρμόνισης ε, της ενοποιημένης φορολογικής βάσης για εταιρεία στο εγγράφο του Ελάν Λαμασούρ. Γίνεται απόπειρα να καλευθεί και η ψηφιακή φορολόγηση στον τομέα της εταιρικής φορολόγησης. Δύσκολο εγχείρημα. Χρειάζεται η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλουμε να καταστούν αυτά λειτουργικά. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερωτηματικό. Είτε θα είναι ξεχωριστή η φορολόγηση του ψηφιακού τομέα ή θα καλύψει η εταιρική φορολόγηση και τον ψηφιακό τομέα. Και στη συνέχεια, το πιο ευαίσθητο θέμα νομίζω είναι το πώς θα καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, πώς θα εισαχθεί περιβαλλοντική φορολόγηση. Εδώ έχουμε μία απόπειρα να γίνει ουδέτερη κατάσταση. Γιατί αν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που α, πάρα αυτά κάποιες χώρες πληχθούν από την φορολόγηση αυτή, ουσιαστικά σκοτώνουμε την πρόταση αυτή εν τη γενέση της. Όπως έγινε και με την ενεργειακή φορολόγηση και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 για τη φορολόγηση ε, των εκπομπών που δεν υπάγονται στο σύστημα ETS ε, ε Αν θέλουμε λοιπόν μια πιο ουδέτερη πρόταση, θα λέγαμε σε ό,τι αφορά τον φόρο άνθρακα στι συζητήσει του 2007 ο πρόεδρο Σαρκόζη ήταν ο πρώτος ο οποίος πρότεινε προσαρμογή του άνθρακα. Μπορεί να το, καλέσουμε να το αποκαλέσουμε αυτό προστασία του περιβάλλοντος κατά του dumping. Υπάρχουν διάφοροι φόροι για το περιβάλλον Όλα αυτά για τις εισαγωγές χωρών, από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν συστήματα εμπορίας ρήπων, ETS. Αυτό θα ήταν, αν θέλετε, ένας πράσινος προστατευτισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προστατευτούμε από το περιβαλλοντικό dumping. Φυσικά, αντιλαμβάνομαι απόλυτα, ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από τις άλλες χώρες να προσθέσω το εξή. Πρόκειται για ένα σύστημα με διάφορε διορθώσει και επιστροφέ. Αν θέλουμε να μην υπάρξουν επιστροφές, θα προτείνουμε ίδιους πόρους με άμεση αποζημίωση για πολλά κράτη-μέλη και να μην ξεχάσουμε αυτή τη φορά και τα λοιπά έσοδα, όπως αποκαλούνται, Κάποια είναι προβλέψιμα, κάποια είναι απρόβλεπτα και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο αποθηματικό. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Lewandowski. Merci pour cette contribution et euh, je donne la parole. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Έτιγκερ να ακούσουμε τις δικές του αντιδράσεις, τις δικές του παρατηρήσεις στα όσα μόλις άκουσε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, τέσσερις εισηγητές και να δηλώσω τον σεβασμό μου. Γιατί τα σχέδια τα οποία προετοίμασαν μαζί με τους βοηθούς τους και τη ε, βοήθεια των ε, τεχνικών επιτροπών. Διάβασα λοιπόν τις, τα κείμενα αυτά και πιστεύω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καθοριστική και σωστή βάση. Και είμαι ευγνώμων που το Κοινοβούλιο αποφάσισε να τα κοιτάξει αυτά με επιτυχημένο τρόπο, προκειμένου το Φεβρουάριο να ληφθούν οι αποφάσεις ε, στις επιτροπές και το Μάρτιο να περάσει στην Ολομέλεια το θέμα. Και έτσι λοιπόν ε, με την ε, γνωμοδότησή σας νομίζω ότι τοποθετήσετε τη σωστή χρονική στιγμή στη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα δημοσιευτεί τον Μάιο, θα ήθελα να σα πω ότι θα προσπαθήσουμε και θα θέλαμε να έχουμε και να συμπεριλαμβάνουμε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο πιο πολλέ από τι δικέ σα προτάσει και τι δικέ σα ιδέε. Η δική μα λοιπόν δουλειά είναι η εξή. Πριν από δύο εβδομάδε έγινε στο Σώμα των Επιτρόπων μια μεγάλη συζήτηση για να τεθούν οι κατευθυντήριε γραμμέ σε μια διάσκεψη με χίλιου περίπου συμμετέχοντε και συμμετείχαν και πάρα πολλοί ε, βουλευτέ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Αρτουή, ο οποίο συμμετείχε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να, να συμπεριλάβουμε όλους τους παράγοντες τους οποίους χρειαζόμαστε και θα μεταβώ και σε δύο πρωτεύουσε προκειμένου να συνομιλήσω με τους αρμόδιους υπουργούς καθώς και με τις επιτροπές των κοινοβουλίων. Τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν κάθε μέρα θα ενισχύουμε τις απόψεις μας μετά από την συλλογή πληροφοριών. Τα πράγματα όμως ακόμα είναι ρευστά από την ε, Σύνοδο των Ηγετών, από την ε, Ανεπίσημο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 ε, Φεβρουαρίου, θα θέλαμε ένα σαφές, μια, σαφής, μια σαφή ένδειξη για το κατά πόσον υπάρχουν προτεραιότητες σε ό,τι αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο πρόεδρος τους και είναι στενές επαφές και ο σκοπός του είναι στις μετέπειτε εργασίες του για το Συμβούλιο για το 2018 και το 2019 να υπάρχει η απαραίτητη ένταση εργασίας σε ό,τι αφορά τις διαβούλευσεις. Έχουμε και κάποια σημαντικά θέματα περιεχομένου επί των οποίων θα καλυφθούμε να αποφασίσουμε. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θέλει να υπάρχει ένα ε, συνεκτικό, ομοιογενές ε, πλαίσιο προπολογισμού για τις 27 χώρες και όχι για ένα διτό σύστημα με, για ευρωζώνη. Και γι' αυτό γιατί. Γιατί μεταξύ των, ε, της Ευρωζώνης και των υπόλοιπων χωρών υπάρχουν όλο και πιο λίγες διάφορες. Ο προπολογισμό για, το 2000, για την Ευρωζώνη είχε προταθεί το 2011 για πρώτη φορά. Τώρα όμως έχουμε 19 χώρες πλέον στην Ευρωζώνη και κατά τη διάρκεια του επόμενου πουδουπού, τα επόμενα λοιπόν 7 χρόνια, θα προσταθούν μία, δύο, ενδεχομένως και τρεις χώρες στην Ευρωζώνη, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί. Θα έχουν γίνει λοιπόν μέλη της Ευρωζώνης. Άρα θα είναι λίγες οι υπόλοιπε χώρες. Θα είναι όλο και πιο λίγε οι χώρε που αποκλείονται. Και έτσι λοιπόν τα πράγματα θα δυσκολεύουν όλο και πιο πολύ για αυτούς ε, επιπροσθέτω δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να υποβάλουμε ένα φιλόδοξο προπολογισμό για τις 27 χώρες και μετά για την Ευρωζώνη να προσθέσουμε άλλες επιπλέον ποσοστίες μονάδες σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ. Ο Μακρόν δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνει στην ε, Βιέννη και σε άλλες χώρες και να μην έχει περιθώρια πλέον. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ισχυρό προπολογισμό για την Ευρώπη των 27. Ε, Υπάρχουν λοιπόν και κάποια κενά φυσικά. Έχουμε το κενό του Brexit καταρχά. Ε, είναι όλο και πιο σαφέ ε, το τι θα γίνει με τους Βρετάνους το 2019, το 2020, στη μεταβατική φάση και μετά το 2020, γιατί προτίθεται να πληρώνουν. Αλλά διαρθωτικά, τουλάχιστον στο επόμενο μισή του Πουδουπού θα μας λείπουν 12 ε, έως 14 δις ευρώ. Θα λείψουν. Δεν πιστεύω λοιπόν ε, καλύτερη ισορροπία από το να πούμε ότι αυτό το κοινό του Brexit θα το κλείσουμε με 50% αναδιαρθρώσεις, εσωτερικές αναδιαρθρώσεις στις ήδη φυστάμενες ε, δομές και 50% με νέα μέσα από τις 27 χώρες μέλη και θα έχουμε και φυσικά το κενό που θα προκύψει και στα καθήκοντα αλλά και στα, στις Γιατί θα υπάρχουν πολλές ακόμα καινούργιε δαπάνες, ε, πολλά καινούργια καθήκοντα, συγγνώμη, αμα, όπου πολλά πράγματα βγάζουν νόημα σήμερα, αλλά δεν είχαν ληφθεί υπόψη το 2013. Δεν ήταν δυνατόν να προβληθούν τότε. Προστασία των σύνορων, για παράδειγμα πολέμηση της τρομοκρατίας, η μετανάστευση, αρρωγή προς τους πρόσφυγες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ενισχυμένη α, αναπτυξιακή βοήθεια, έρευνα για την άμυνα, άμυνα. Σε όλα λοιπόν τα ζητήματα αυτά ε, είναι σαφής η προστιθεμένη αξία. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένα τα κράτη μας έχουν 100.000 ε, συνοριακούς ε, συνοριοφυλακές στα πλαίσια της Frontex. Δεν χρειαζόμαστε να είμαστε μαθηματικοί για να δείξουμε ότι καλύτερα θα ήταν να είναι σωστή και χωρίς χάσματα, χωρίς κενά η συνοριακή φύλαξη, όλοι να καταχωρίζονται και να προωθούνται. Μετά να αποφασίζεται κατά πόσο θα ενσωματωθούν στι κοινωνίε μας ή θα επιστραφούν. Αντιστρόφως όμως, σε ό,τι αφορά τα ιστορικά ευρωπαϊκά σύνορα, να διατηρηθεί και να ανακτηθεί η πλήρης ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ και στη Γερμανία ε, και Δανία. Η έλεγχη των σύνορων είναι πιο αυστηρή παρά ποτέ. Αυτό δεν πιστεύω ότι είναι πιστικό μεταξύ της Αυστρίας και Γερμανίας. Η έλεγχη είναι πιο αυστηρή παρά ποτέ. Και αυτό πραγματικά δεν θεωρώ ότι έχει νόημα στη Βαβαρία, οι φίλοι από το κόμμα μου, αν θα θέλαν να κάνουν τέτοιου συναριακούς ελέγχου, ε, το οποίο δεν γίνεται φυσικά από πλευρά ε, συνταγματικού δικαίου, γιατί αυτό αποφασίζεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αγαπητοί φίλοι, αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τις εκλογές σε επίπεδο ομοσπονδιακών κρατηδίων. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσον το Κοινοβούλιο θα ακολουθούσε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα επόμενα χρόνια να αυξήσουμε τις θέσεις στη στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Βούλγαρια, Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία να συγχρηματοποτήσουμε ε, την αύξηση των θέσεων αυτών. Γιατί από μόνες τους δεν πρόκειται να το καταφέρουν προκειμένου να έχουμε ε, μια σωστή πλήρη προστασία των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Γιατί αν δεν υπάρχει τέτοια προθυμία, τέτοια θέληση, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα σύνορα και να ανακτήσουμε την πλήρη ελεύθερη κυκλοφορία, την πλήρη κατάργηση των εσωτερικών συνόρων. Αυτό θα ήταν πραγματικά μια μεγάλη κίνηση για το που και όχι απλά να αυξηθούν κατά 150 θέσεις στη Frontex ε, οι συνοριοφυλακέ. Είμαστε επιτεθειμένοι λοιπόν να εγγυηθούμε την πλήρη ελεύθερη μετακίνηση στις 27 χώρες και να υπάρχει πλήρης 100% ε, αδιάτρητη προστασία των εξωτερικών συνόρων. Δεν θέλω λοιπόν να εξαιρέσω προγράμματα περικοπών. Όχι. Αυτό θα ήταν ε, μη έντιμο στην ε, συνοχή, στη γεωργική πολιτική, χωρίς σημαντική πρικοπή, που ωστόσο δεν θα βλάψει τα προγράμματα, δεν θα τα βγάλουμε πέρια. Και θα ήθελα να εξαιρέσω δύο προγράμματα, Erasmus Plus και τον Ορίζοντα Ευρώπη, έρευνα, ανάπτυξη και νεολαία. Και θα ήθελα να πω το εξή. Τα προγράμματα όπου υπάρχει σημαντική προστιθέμενη αξία. Χθε ήμουν σε μια μεγάλη διάσκεψη όπου ήταν και ο συνάδελφος ε, Αρτουή και τα ε, ο Αλληλέος ε, ή τα διαστημικά προγράμματα. Και όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέονται με αυτό, αυτά γίνονται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να περικόψουμε εδώ τα μέσα. Μη σας πω ότι χρειάζεται και σημαντική αύξηση. Περικοπές στα προγράμματα πολλαπλών προ, παραγόντων και να μην υπάρχει περικοπή σε κάποια επιλεγμένα λίγα προγράμματα. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για το θέμα των ανώτατων ορίων, των ανοφλίων. Θεωρώ ότι αυτά που αναφέρετε είναι σκόπιμα και φιλόδοξα. Εδώ, αν ήμουν βουλευτής, το ίδιο θα έκανα. Την ίδια πρόταση θα κατέφετα. Αντιστρόφως όμως θα πρέπει να σα πω από τι υπηρεσιακές μου επισκέψει ότι υπάρχουν κάποια κρατημέλη Δεν μιλάμε για καθήκοντα, για δαπάνες, απλά λέμε ότι πολύ ωραία 1,0%. Γιατί αλλιώς δεν θα συμφωνήσει το Συμβούλιο. Κάποια κρατημέλη λοιπόν αυτό ισχυρίζονται. Νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε μία σειρά από κρατημέλη για να κάνουν καλύτερες δαπάνες σε ό,τι αφορά το 1,0% στο τρέχον που δουπού. Αυτό το 1,0% ε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών μας και θα πρέπει να έχουμε διάφορα άλλα ζητήματα που όπως για παράδειγμα η μετανάστευση, η άμυνα, η προστασία των συνόρων, αυτό όλα δεν μπορούμε να τα καλύψουμε αυτό το 1%. Θα πρέπει λοιπόν να καταργήσουμε αυτή την ε, ε, ανταγωνισμό μεταξύ της άμυνας και της γεωργίας, για παράδειγμα, μεταξύ της ε, μετανάστευσης και της ασφάλειας. Γιατί όλα αυτά θα ήταν ενδυνάμει διχασμοί της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Εμείς είμαστε στο 1,1 χ. Δηλαδή κατά ελάχιστο όριο 1,1 ε, κατά ανώτατο όριο 1,2%. Αυτή τη μετακίνηση τη θεωρώ απαραίτητη. Και να σας πω και κάτι άλλο Έχουμε και το πακέτο της 6ης Δεκεμβρίου με τα νέα μέσα για την προενταξιακή βοήθεια για την Ευρωζώνη, για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων, για τις θέσεις εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε μεγαλύτερες προσαρμογές στο 1,2 από ότι στο 1,1%. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Θα ήθελα να ενσωματώσουμε την Ευρωπαϊκή Ενεπταξική Βοήθεια, να τη βάλουμε στον προπολογισμό. Θεωρώ ότι αυτό θα ανταποκρινόταν και στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου για να είναι μια μόνιμη εργασία και η οποία θα ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αυτό εξαρτάται από το 1,0, 1,1 ή 1,2%. Ένα τρίτο παράδειγμα, για παράδειγμα. Και την πλήρη δυνατότητα μεταφορά των μη δαπανόμενων πόρων να είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο δεύτερο τέταρτο έτος. Με το 1,2% λοιπόν μπορούν να επιτευχθούν τέτοιες ε, προτεραιότητες που θα έχουμε θέσει και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην κυρία Τωμά για το γεγονός ότι δέχεται για μία φορά ακόμα τα 7 έτη, γιατί αν έχουμε την θητεία της Επιτροπής 5 έτη, του Κοινοβουλίου 5 έτη, η... αν θέλουμε να φτάσουμε στο 5 συν 5 χρόνια, δεν είναι δυνατόν να κοινοβούλιο την τελευταία χρονιά και μια θητεία, μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία επίση χρονιά τη θητεία σα να καθορίσουν την επόμενη αμα, ισχύ του που, τα επτά χρόνια είναι η σωστή λύση ω μεταβατική λύση. Και αυτό χαίρομαι που μπορώ να το ανακοινώσω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για την ρεσιμότητα. Η οικονομική ρεσιμότητα ή την ρεσιμότητα για το κράτος δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν οι νομικοί μας ε, να φροντίσουμε να έχουν όλες τις τεχνικές ε, και νομικές ε, διατάξεις. Το πρώτο τελευταίο σημείο. Headings. Τα κεφάλαια αποτελούν πολιτική. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν σε ή σε 7 κεφάλαια να μεταβούμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ασφάλεια και άμυνα. Ένα κεφάλαιο για παράδειγμα. Ένα άλλο κεφάλαιο θα μπορούσε να είναι καινοτομία, μέλλον, νέα γενιά. Προκειμένου να κάνουμε πιο ξεκάθαρο στους πολίτες και στους φορολογούμενους σε τι επενδύουμε, πού βρίσκεται η προστιθέμενη αξία για τον κόσμο στην Ευρώπη. Ακόμα, ακόμα για να γίνουν τα κεφάλαια πιο σαφή για τον Ευρωπαίο πολίτη. Να μην ξέρουν δηλαδή μόνο οι τεχνικοί και περιογνώμονε τι είναι το 1β1α και το καθεξή. Τελευταίο σημείο, επιτρέψτε μου. Το Μάιο θα προτείνουμε το έκτο πουδουπού. Πρώτο ήταν το Ζακτελόρ, το 88. Αλλά ω τώρα, μέχρι και το πέμπτο πουδουπού, δεν υπήρχε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο. Μετά Δεν η κατάσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλην τη θέση σε ισχύ το 2021 θα υπάρξουν ευρωεκλογέ. Αυτό δεν έχει παρουσιαστεί ως φαινόμενο ω τώρα και αυτό αποτελεί μεγάλο κίνδυνο. μεσολαβούν ευρωεκλογέ. Γι' αυτό λοιπόν ε, το χειρότερο σενάριο θα ήταν για μένα το εξή. Να υποβάλουμε την πρόταση να γίνει ο προεκλογικό αγώνα και εσεί να κάνετε προεκλογικό αγώνα και κάποιοι να υποσχεθούν ναι, παράδεισο στην Ευρώπη με πολλά χρήματα. Άλλοι να βγουν να πούν ότι α, όχι, δεν θα δώσουμε στου γραφειοκράτε τη ε, Βρυξέλλε ε, χρήματα. Και θεωρώ ότι αυτό μπορούν να το κάνουν οι κορυφαίοι υποψήφοι. Μετά θα προκύψει ένα καινούργιο κοινοβούλιο, θα συσταθεί ένα νέο ευρωκοινοβούλιο, θα υπάρχουν εσωτερικέ ε, ε, διαδικασίε για τη σύνθεση των επιτροπών και το καθεξή. Θα γίνουν οι ακροάσει των επιτροπών. Θα συσταθεί το νέο σώμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι νέο ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο ε, θα πρέπει να τηρήσει και να αποτυπώσει ένα τμήμα των δεσμεύσεων των, προεκλογικών στο πουδουπού. Θα έχουμε 20 νέου επιτρόπους και έτσι θα φτάσουμε την άνοιξη του 2020. Και έτσι το Δεκέμβριο του 2020 θα σημειώσουμε τα αποτελέσματά μας και θα, κάνουμε, θα επαναλάβουμε τα παλιά λάθη. Το 2021 σε ό,τι αφορά τη συνοχή, την έρευνα για πολλά προγράμματα θα είναι μια χαμένη χρονιά, όπως ήταν χαμένη χρονιά το 2014. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε τώρα, αλλά μπορούμε να έχουμε τη φιλοδοξία. Σας ευχαριστώ που έχετε και εσείς την φιλοδοξία για να κάνουμε μια απόπειρα από τον Μάιο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 να το δούμε αυτό ως προτεραιότητά μας και εσείς και εμείς και ελπίζουμε να το δεχτείτε και το Συμβούλιο. Και να μην τα αναβάλουμε όλα αυτά διαρκώς και να θέσουμε ένα μήνυμα ότι τη στιγμή που οι Βρετανοί φεύγουν με όλες τι διαφορέ που έχει το Κοινοβούλιο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό σημάδι καλή διακυβέρνηση. Α το προσπαθήσουμε. Είναι λίγο δύσκολο, δεν λέω. Αλλά το να μην το προσπαθήσουμε καν θεωρώ ότι θα ήταν πραγματικά ε, κάτι το οποίο θα μα απογοήτευε και θα έπρεπε να προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ. Είναι από ό,τι βλέπετε πολύ στρατευμένος ο Επίτροπος στην προετοιμασία του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και θέλει να χαρακτηρίζεται από μια ευρωπαϊκή φιλοδοξία που να ανταποκρίνεται και αυτή στις προσδοκίες των πολιτών για μια Ευρώπη του μέλλοντος και μια Ευρώπη που προστατεύει. Ε, δεν μιλήσατε για τους ίδιους πόρους ιδιαίτερα. Θέλετε να μας ε, ενημερώσετε λίγο περισσότερο. Μόνο για σαφέ ότι αν ε, δεν το αναφέραμε αυτό στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δουλειά του Μάριο Μόντι και των υπόλοιπων τη ομάδα υψηλού επίπεδου θα πήγαινε στα σκουπίδια. Είναι σαφέ οι προσδοκίε σα. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε και νέε προτάσει και περαιτέρω προτάσει. Ένα τμήμα των προτάσεων δε αυτό που είναι ενδιαφέρον ε, στις ίδιου πόρους. Υπάρχουν ε, κάποιοι οι οποίοι είναι γενικά κατά. Δεν το θέλουν. Θέλουν το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 100% αν γίνεται να εξαρτώνται από τις εθελοντικές δαπάνες των κρατών μελών. Τι. Ο φόρος ε, κύκλου εργασιών θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, να να Και θέλουμε δύο-τρεις προτάσεις και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Λεβαντόφσκι και του υπόλοιπου, να ε, ε, ενσωματωθούν. Αυτό ωστόσο που λείπει είναι το εξή. Ακόμα παρακαλέσω, ακόμα και αν έχετε αμφιβολία για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα των ιδίων πόρων, αν ο καθένα ε, αρχίσει και εκφράζει τι αμφιβολίε του και δεν συμφωνεί με το ένα και με το άλλο, θα πάει στραβά όλο το σύστημα. Νομίζω ότι η μεταφορά των εσόδων του ETS αποτελεί αποτελεί κάτι εύκολο, ένα εύκολο φόρο σε ό,τι αφορά και για την ε, αποδοχή των ευρωπαϊκών φόρων από τα εθνικά κρατημέλη, σε ό,τι αφορά τους ε, ευρωπαϊκούς στόχους, για παράδειγμα, για τη μείωση των εκπομπών. Είναι ευρωπαϊκή στόχη αυτή, με σαφή ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Στο θέμα της προστασίας του κλίματος έχουμε μια αξιοπιστία να επιδείξουμε. Ε, το σύστημα λοιπόν ETS και η εμπορία των φόρων αυτών αποτελεί δική σας νομοθεσία όλα είναι ευρωπαϊκά. Μόνο από τα έσοδα πηγαίνουν στους ε, εθνικού προπολογισμού. Άρα τον να με την ε, ζωή του κύριου Λεβαντόφσκη πιο εύκολη όταν πηγαίνει στη Βαρσοβία. Σε ό,τι αφορά του στόχους της μείωσης, ε, αν Το θέμα των χρηματοοικονομικών αγορών το κοιτάμε με πολύ ενδιαφέρον για τις ΕΚΤ να έχουμε πολύ σημαντικά έσοδα, τα οποία θα βοηθήσουν πολύ τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τρίτον, Ακούλε οι οποίες δεν μπορούν να ανακυκλωθούν και να τερματιστούν οι εξαγωγές προς την Κίνα κτλ. Φόροι να υπάρχουν, οι οποίοι θα, είναι νόη, θα έχουν νόημα μόνο αν γίνουν με μη γραφειοκρατικό τρόπο. Να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να έχουμε να κάνουμε με τις πρώτες θα έχουμε να κάνουμε με το προϊόν της πλαστικής σακούλας του Καρφούρ, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω ότι Δύο-τρει προτάσει σα θα τι συμπεριλάβουμε στην πλευρά των εσόδων και θα προσπαθήσουμε όντω σε επίπεδο υψηλού επίπεδου να έχουμε μια ομάδα εκπροσώπων. Δεν είχαμε πετύχει τίποτα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν θα αντικατόπτριζε μια πολύ υψηλή ποιότητα δουλειά ε, η οποία έγινε στο, στην ομάδα υψηλού επίπεδου και από του συζητητέ. Ε, Ευχαριστώ κύριε θα δώσω καταρχήν το λόγο στους σκιώδεις ηγητές. Ένας σκιώδης εισηγητής ανά ομάδα. Και για τα δύο ζητήματα. Πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ήδη Μετά θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές ε, για τις... Ε, θα μιλάνε έτσι. Οκ. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Θα ήθελα να πω Η εργασία των εισηγητών θεωρώ ότι είναι ευρία πλειοψηφία. Δεύτερον, έχουμε την αποφασιστικότητα του Επιτρόπου. Πάρα πολύ θετικό, του ΑΕΠ για τον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι ρεαλιστική πρόταση. Και μάλιστα θα έπρεπε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα της διαπραχθή η πολιτική μας φιλοδοξία και οι προτεραιότητες μας το αντίθετο. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι ως 27 είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε σύλλογοι. Οι πολιτικές που λειτουργούν θα πρέπει να διατηρηθούν. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Οι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει, οι καινούριες προτεραιότητες θα πρέπει να ε, πρικοδοτηθούν με καινούριου πόρους. νησιν 3 ισχύει, οπότε μέχρι το 2023 θα έχουμε εκεί προπολογισμού. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε γρήγορα. Έχετε τρία λεπτά, αλλά μιας και προεδρεύω εγώ δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, λέω κύριο Βιώτη, ευχαριστώ τον Επίτροπο Έτεγκερ για τη συζήτηση σήμερα το πρωί, γιατί μα επιτρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάπω τι ιδέες μας για τη δουλειά την οποία έχουν κάνει μέχρι τώρα οι εισηγητέ για τα δύο έγγραφα. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε λίγα θέματα, ιδιαίτερα στο θέμα του επόμενου ε, δημοσιονομικού πλαισίου γιατί εδώ θα έλεγε εκπροσωπείται στο άλλο θέμα μάλλον και η πολιτική μας θέση σαν ομάδα από την κυρία Τομά. Ε, για το πολιετές δημοσιονομικό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι η φιλοδοξία στην οποία όλοι έχουμε, την οποία, στην οποία όλοι προσβλέπουμε, να μην περιμένουμε το τέλος του 2019 για να κλείσουμε εμπασπετός το θέμα, αλλά να τελειώσουμε πριν από τις ευρωεκλογέ. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μετατραπεί σε κάτι το οποίο θα μειώσει τα πάντα, θα περικόψει τα πάντα. Βέβαια ε, πάντα στους, ε, όταν εξετάζουμε τους προϋπολογισμούς υπάρχει ένα τελικό χρονικό όριο πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να πάμε και μέσα στο περιορισμένο αυτό χρονικό πλαίσιο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη δημοσιονομική διαδικασία. Η φιλοδοξία μας εδώ είναι από τη μία να συνδυάσουμε ισχυρές πολιτικές και αντίστοιχους πόρους που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτικών αυτών. Στο θέμα των ιδίων πόρων τώρα ε, θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Το θέμα το ψηφιακό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, διότι τα κράτη-μέλη δεν καταφέρνουν από μόνα τους να τα αντιμετωπίσουν. Και εγώ δεν θα ήθελα το Facebook να αποφασίζει το πώς πληρώνω και πότε ε, και πόσα, όπως είχε πει ο ιδρυτής του Facebook πριν λίγο καιρό. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει τι φόρους θα πληρώνουν ή ε, ψηφιακή πάροχη. Δεύτερο θέμα για την ε, φορολογία του οικολογικού τύπου. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε είναι τα ε, φορολογικά dumping και τα δημοσιονομικά dumping στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εισάγουμε ένα νέο φόρο. Και επίσης δεν θα πρέπει να δημιουργούμε σε επίπεδο περιβαλλοντικό ε, τέτοιου είδους οικονομικά ντάμπινγκ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όχι να θέλουν βέβαια οι επενδυτές να πάνε στο εξωτερικό γιατί έχουν ε, φορολογικές διευκολύνσεις περισσότερες. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Επιτροπέ. Θα μιλήσω για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πόρους θα πρέπει να δαπανούνται αποτελεσματικά. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι οι πληρωμές θα δαπανούνται με εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΕΚ και από την εισφορά των κατανομέλων. Κατά δεύτερον, το νέο σύστημα θα πρέπει να εστιάζεται σε τομείς που οι ωφέλη, οι δαπάνες θα πρέπει να εστιάζονται σε project τα οποία θα είναι ε, δυνατά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και όχι τόσο σε κανόνες σε ό,τι αφορά την ταπάνη των πόρων για μεγαλύτερη διαφάνεια. Και θα πρέπει να την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και την ευρωπαϊκή προβολή, αν θέλετε. Ευχαριστώ από τους πράσινους. Έχουμε δύο και γραμμένους. Πρέπει να επιλέξετε όμως έναν. Ποιος θέλει να αποφασίσει η πρόεδρος, μήπως η συντονίστρια ποιο θα μιλήσει από... Α, συγγνώμη, λέει ο προεδρό Μαδάμ Ελπίζω να είμαι πιο σύντομη. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια προσέγγιση η οποία θα έχει κάποιες βασικές αρχές. Μείωση ανεργίας, μείωση των διαφορών σε περιφερειακό και τοπικό και εθνικό επίπεδο και προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις σε βάση αλληλεγγύη, σε βάση βιώσιμης ανάπτυξη. Αν δεν συμφωνήσουμε γι' αυτά, θα συμβάλλουμε στον κατακαιρματισμό και στις συγκρούσεις. Και αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον, κύριε Πετρόπε, είναι αυτό που είπατε για τον διχασμό της ευρωπαϊκής οικογένειας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αν αυξήσουμε τις ε, δαπάνες ε, στην ε, άμυνα και δημιουργήσουμε το φρούριο της Ευρώπης, θα... Το έχουμε δει και στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία, με τα σύνορα, τα σκληρά αυτά σύνορα. Νομίζω ότι η οικογένεια ευρωπαϊκή μπορεί να ωφεληθεί από τα διδάγματα του παρελθόντος, προκειμένου να μην αυξήσουμε αυτή την αίσθηση της αρέσκειας και φόβου στην Ευρώπη και πιστεύουμε ότι οι μεγαλύτερες δαπάνες στα στρατιωτικά ζητήματα και η μείωση ε, στις δαπάνες για την κοινωνική ανισότητα, για την ε, ανεργία είναι ανησυχητική. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό ισοσκελισμό και να υπάρχει και αλληλεγγύη μεταξύ των 28 κρατών μελών. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι κοινωνικέ πολιτικέ, την εκπαίδευση, την έρευνα, την κατάρτιση, την υγεία, ενσωμάτωση, απασχόληση και απλές πολιτικές για την φορολόγηση και φυσικά καταπολέμηση και των φορολογικών παραδείσων. Θα πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στις συντριπτικές αρχές της Ένωσης, αλληλεγγύη, μια κοινωνική Ευρώπη για τον κόσμο. Αυτό ζητάνε λοιπόν όλοι. Ε, προσβλέπω λοιπόν στη συνέχιση της συζήτησης και ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Νομίζω ότι ήμουν και πιο σύντομη και αξίζω το βραβείο. Ναι, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, κύριε Τριέτα, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Τρούπερ, και μια και είσαστε και εισηγήτρια από. Θα μιλήσω στα αγγλικά και μετά θα μιλήσω γερμανικά. Είναι η τρίτη φορά λοιπόν που συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πουδοπού και φαντάζομαι ότι οι συγκρούσεις θα είναι ακόμα πιο δύσκολε. Ε, σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, γιατί οι διαφορές μεταξύ των χωρών που είναι καθαροί φορές είναι ακόμα μεγαλύτερες και κοιτώντα και σε επίπεδο του Βυσσιακράτη νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αυξηθεί με τις χώρες αυτές ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό. Συμφωνώ και με τον κύριο και με του συζητητές με το φιλόδοξο στόχο του 1,3%. Συμφωνώ και ήμουν πολύ απογοητευμένη όταν ο Μάρτιν Σούλτ την τελευταία φορά ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησε να μειωθεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό για πρώτη φορά. Ήταν κακό αυτό, κακό ω προηγούμενο. Εμεί ω πράσινοι δεν συμφωνήσαμε και νομίζω ότι τα τελευταία 3-3,5 χρόνια καταδεικνύουν ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό για την διαχείριση των συνόρων, την έρευνα, την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, ε, την εκπαίδευση, ε, σταθεροποίηση των αφρικανικών χώρων, προκειμένου να μην φεύγουν τόσο πολλοί πρόσφυγες από τις χώρες αυτές και τα δεικνύουν ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και τώρα να μιλήσω γερμανικά. Συμφωνώ λοιπόν με την προσέγγιση του Επιτροπού Ρότινγκερ ότι θα πρέπει να γίνουν σημαντικές, ε, κάποιες μάλλον στοχευμένε ε, μειώσει σε σημαντικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Συνοχή, το Γεωργικό Ταμείο. Εγώ ω στα μεγάλα στους ομίλους. Αυτό δεν είναι κάτι το βιώσιμα. Και δεν πρόκειται. Αυτά τι παρεσίου θα πρέπει να αποτυπωθούν στο επόμενο που Και αυτό Λοιπόν, θεωρώ ότι αποτυπώνεται και στην πρόταση του κυρίου Όλμπριχτ και στα αποτελέσματα του Παρισιού στο νέο Πουδουπού, θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να οδεύουμε προς την καταστροφή του πλανήτη. Κοιτάξτε τι γίνεται με τα αποτελέσματα του Παρισιού στο νέο Πουδουπού, θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να οδεύουμε προς την καταστροφή του πλανήτη. Κοιτάξτε τι γίνεται με τις ε, πλημμύρες, με τις πλημμύρες ε, λάσπη στην Καλιφόρνια, έχουμε όλο και πιο πολύ ξηρασία, περίμωση. Επίση, συμφωνώ με τον Επιτροπό του Έτογκερ ότι δεν χρειαζόμαστε προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Όχι, θα πρέπει να έχουμε πιο υψηλό ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα πρέπει να συμφωνούν, να συμμετέχουν όλοι. Και θα πρέπει σιγά σιγά να προσταθούν και οι υπόλοιποι στο ευρώ, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντική πολιτική να υπάρχει. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκέ δυνάμει, όχι για να κάνουμε ευρωπαϊκή επίθεση, για να αναλάβουμε τι παγκόσμιε ευθύνε μα και κυρίω να ενώσουμε τι δαπάνε μα αυτέ και να μην έχουμε ξεχωριστέ δαπάνε και να μην εξαρτώμαστε και από τους Αμερικανούς. Υποστηρίξουμε, ναι, αν θα θέλετε πάρα πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να φύγει ο επίτροπο και θα ήθελα να πάρει το λόγο ο κ. Ζαλή. Σα είχα δώσει ένα λεπτό μόνο το λόγο. μεγαλύτερη σημασία λοιπόν στην ε, ναι, διακόπτει ο πρόεδρο. Σα παρακαλώ, αν θα θέλετε μετά, αφού φύγει ο επιτροπό, έχετε το λόγο, αλλά σύντομα. <clears throat> Θα είμαι πολύ σύντομο. Καταρχά, για το πολιετέ δημοσιονομικό δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειε, και ο κ. Τζάνι. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για τον γενικό στόχο. Σήμερα το πολιετέ δημοσιονομικό παρουσιάζει μία πρόκληση ιδιαίτερα για τις χώρες οι οποίοι είναι καθαρείς φορείς. Με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, η διαφορά ανάμεσα στα χρήματα τα οποία αποδίδονται και στα χρήματα τα οποία λαμβάνονται θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό επηρεάζει την Ιταλία, τη Γαλλία και θα επηρεάσει αρνητικά τον προϋπολογισμό των χωρών αυτών. Γι' αυτό θα πρέπει και η Επιτροπή μας και τα κοινοτικά όργανα θα πρέπει να μην αλλάξει η διαφορά ανάμεσα στα χρήματα που δίδονται και σε αυτά που λαμβάνονται, μειώνοντας κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν είναι παραγωγικές και αυξάνοντας ίσως κάποιες θέσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες έχει αποδείξει το παρελθόν ότι είναι αποτελεσματικές. Είναι μια πολιτική συζήτηση. Υπάρχει χώρος, αυτό το είδαμε και στη συζήτηση για την προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία και είδαμε ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση βρίσκονται λύσεις. Τώρα για τους ιδίους πόρους. Και εδώ διάβασα την έκθεση των δύο εισηγητών και έχω πάρα πολλές αμφιβολίες. Δεν βλέπω κάποια καινοτόμα στοιχεία η αναζήτηση των ιδίων πόρων στην ουσία ε, δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε παρά μόνο με νέους φόρους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το roaming είναι κάτι το οποίο το αποδεικνύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό καταργώντας το roaming, όμως περνούσε στην Ιταλία, είχε προτείνει να υπάρξει φόρος για τις χρηματοπιστωτικές ε, ε, συναλλαγές τα αποτελερνούσε στην Ιταλία, είχε προτείνει να υπάρξει φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Τα αποτελέσματα αυτού του φόρου είναι σαφώς πολύ χαμηλότερα από ό,τι περιμέναμε και σε επίπεδο συνολικών εσόδων και σε επίπεδο εφαρμοστή, οι οποίες κανονικά σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών μεγεθών θα έπρεπε να ενταχθούν στην Ευρωζώνη, με τέτοιου είδους ε, φόρους θα φύγουν από την Ένωση. Οι κίνδυνοι λοιπόν που δημιουργεί ο νέος αυτός φόρος είναι πάρα πολύ υψηλοί. Τώρα σχετικά για τη φορολογία στα κανάλωση του πλαστικού, καλώς. Αν στόχος είναι νέοι πόροι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και τα δύο αυτά σαν στόχοι δεν συνδυάζονται. Ο κύριος Επίτροπος πριν φύγετε να μας μεταφέρετε τις συστάσεις σας. Επιτρέψτε μου να σε τρία σημεία για σήμερα και θα προσπαθήσω σίγουρα να κάνουμε συζητήσεις και στις πολιτικές ομάδες αλλά και στις ε, επιτροπές που γνωμοδοτούν για το ευρωπαϊκό προπολογισμό. Καταρχάς στα ψηφιακά. Δύο σημαντικές πτυχές να τονίσω. Η πρώτη οι επενδύσεις στις ε, ψηφιακές τεχνολογίες, σε ψηφιακές υποδομές, σε ψηφιακή εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως Εφόσον η ψηφιακή εξέλιξη είναι η πιο καθοριστική εξέλιξη, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και ένα κεφάλαιο για τα ψηφιακά προκειμένου να τα ομαδοποιήσουμε όλα αυτά, αλλά και για να επισημάνουμε συμβολικά τη σημασία των ψηφιακών προγραμμάτων στην ευρωπαϊκή αυτή, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεύτερη πτυχή. Οι πλατφόρμες με, που εργάζονται με δεδομένα, πώς ε, έτσι, και ε, ο κινητήρας από το Βουκουρέστι, από την Πρωθυσλάβα, άλλα τμήματα, Οι οι οικονομικοί μας δίκαιοι και εργάζονται απεγνωσμένα. Θα βρούμε λοιπόν έναν τρόπο ο οποίος να είναι αξιόπιστο Όταν δηλαδή οι μεγάλες, οι μεγάλοι όμιλοι έχουν έδρα σε κάποιο φορολογικό μέσα στο έτος. Κατά δεύτερον, στην άμυνα. Το θέμα δεν είναι να έχουμε πιο πολλέ δαπάνε για την άμυνα. Το θέμα είναι να έχουμε πιο αποτελεσματικέ δαπάνε και μπορούμε να αποδείξουμε τιμά από ένα ευρωπαϊκό σύστημα συγχρηματοδότηση. Και άρα στο δημοσιονομικό έτος 2000 μιλάμε για πιο πολλέ δαπάνε, μιλάμε για καλύτερε δαπάνε. Και αυτό που είναι σαφέ, είναι το εξή. ότι αν ε, συντονίσουμε τις προμήθειες και, ε, να κάνουμε τέτοιες ε, διαγωνισμούς με 5 δις. Το πόσα θα δαπανίσουμε είναι άλλο θέμα. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει καλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός. Αυτό είναι σαφές νομίζω και είναι και ξεκάθαρο. Οι Αμερικανοί για ένα δολάριο έχουν πολλά πάνε Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα όπως και ο Αμερικανός. Κυρία Τρίπελε, θα συναντηθούμε και κατηδίαν ε, σε έδωσα κάποιες ώρες ε, και ημερομηνίε και γιατί ό,τι φορά το θέμα των ταινιών και του πολιτισμού μας. Ε, δώσατε κάποιες προτάσεις στα σύμφωνα των όριων, των ε, γεωκτημόνων κτλ. Και από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχουμε μία αξιολόγηση για το κατά πόσον το 20% στο σύνολο του προπολογισμού μπορεί να συνεχίσει να δαπανάται και τα επόμενα χρόνια. Το greening αυτό ήταν επιτυχέ τελικά. Κατά πόσον ε, εγγυάται την ε, ποικιλία, την ε, βιωσιμότητα των ε, εκτάσεων μας. Ενδεχομένως να χρειαζόμαστε καλύτερα, πιο εξελιγμένα εργαλεία από ότι αυτά που έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σας θέσω ένα ερώτημα. Αν συμφωνήσουμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο τον, την άνοιξη του τρέχοντος έτους, αυτό επιτρέπει στην Κομισιόν να εφαρμόσει μια δραστική απλοποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και των διαδικασιών. Γιατί Υπάρχει ένα σοβαρό τον ευρωσκεπτικισμό και την ευρωφοβία. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπέ. Δύο λεπτά ο καθένας. Ο Μαρινέσκου για την Ήτρα και την Τραν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χάρηκα για την δήλωση του, του Επιτρόπου ότι θα στηρίξει την πολιτική για το διάστημα. Το ζητήσαμε χτες και χαίρομαι που θα κρατήσει περισσότερα κονδύλια γι' αυτό. Η πολιτική μεταφορά από την άλλη μεριά ελπίζω ότι θα χρηματοδοτηθεί στο ίδιο επίπεδο με την αρχική πρόταση του Επιτρόπου Λεβαντόφσκι πριν από έξι χρόνια και όχι με περικοπές και όπως αναφέρεται και ε, στην έκθεση Όλμπριχτ και Τόμα ελπίζω ότι ε, και ότι θα υπάρξει αύξηση κατά 50% στην ε, χρηματοδότηση όπως Κύριε Γιάτεν Μάκη για την ένδυ. Θα είμαι σύντομη Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την μετάβαση στην βιωσιμότητα. Η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αναλάβει πολλές διεθνεί δεσμεύσει για το περιβάλλον. Στο προπολογισμό όμως δεν προβλέπεται αρκετή χρηματοδότηση για να ικανοποιηθούν οι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει. Να υλοποιηθούν οι υποχρεώσει μας. Μετά Ακούσαμε πολλές όμορφες αλλά μη ρεαλιστικές ιδέες. Ιδιαίτερα υπό το φως του κενού που θα δημιουργήσει το Brexit. Πόσα... Τι αύξηση χρηματοδότηση μπορούμε πραγματικά να περιμένουμε. Αυτό πρέπει να το δούμε εμείς εδώ ως Κοινοβούλιο. Έγινε αναφορά και στην φορολόγηση. Θα πρέπει να δούμε εναλλακτικές, εναλλακτικά ο κ. Χάουαρθ. Πολιτικές όπως τις συνοχής. Η πολιτική συνοχή όμως εξακολουθεί να είναι η πιο σημαντική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μερικές από τις μεγαλύτερες θα εξακολουθήσει να επιτρέπει τη χρηματοδότηση όλων των περιοχών που το χρειάζονται η περιφέρει με διάμεση αναθεώρηση. Η Επιτροπή επίσης στηρίζει πέρα, να αποδεικνύουν ότι είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. Ε, για τους ίδιους πόρους, ε, ε, αν χρησιμοποιήσουμε ε, ε, φόρος όπως αυτή των πλαστικών ε, ως αντικίνητρο μην περιμένουμε θα έχουμε μεγάλα έσοδα. Από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικός ένας φόρος ψηφιακός. Στις ψηφιακές συναλλαγές αυτό είναι ένας μοντέρνος φόρος. Ένας, να δούμε πόσο θα είναι και ποιο θα είναι. Γιατί η θέση της Βρετανικής κυβέρνησης δεν είναι βιώσιμη και θα πρέπει να πληρώσει η Βρετανία για πρόσβαση στις αγορές που θέλει. Ευχαριστώ. Οι φόροι που αλλάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι φόροι οι οποίοι για την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Επιτροπή ΔΕΒΕ ότι υπάρχει η αξίωση για 0,7% ε, του ΑΕΠ του Ευρωπαϊκού Συναπτυξιακή Πολιτική. Προωθήσουμε στον υπαριθμό 2 Έχουμε την ψυχική ασφάλεια και την ασφάλεια τροφίμων. Στο νούμερο 6 έχουμε το καθαρό νερό. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να φροντίσουμε να έχουμε μια προληπτική ε, προσέγγιση και να σκέφτονται στη διοίκηση όλων αυτών των δομών. Πολλά χρήματα χάνονται σε φορολογικού παραδείσου και έχουμε και ε, μια έκθεση του Ρεκτικού συνεδρίου που καταδεικνύει μέσα αφήνεται στοιχεία σήμερα και νομίζω ότι λίγο πολύ όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες... Έχουμε να κάνουμε με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και την προστιθέμενη αξία. Οι προτεραιότητες είναι προστιθέμενη αξία. Έχουμε νέες προτεραιότητες όπως η μετανάστευση, η άμυνα, η ασφάλεια. Έχουμε παλιές προτεραιότητες. Πώς τώρα η προστιθέμενη αξία μπορεί να επιτευχθεί έρευνα, αμυντικές προμήθειες. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη συνοχή με κάποιο νέο τρόπο, να υπάρξουν νέες ιδέες, ας ξεχάσουμε τις παλιές δομές πολιετούς δημοσιονομικού. Και τώρα για τους ιδίους πόρους δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να ε, εισάγουμε έναν ο κόσμος δεν θέλει ένα κατάλογο περίπλοκων φόρων που προέρχεται από τις Βρυξέλλες. Ας στοχεύσουμε κάτι των πολιτικών, γιατί νομίζω ότι ο Επιτρόπος έχει σκοπό τα μέτρα των γεωργικά να αναπευθούν ε, σε μεγάλο βαθμό στο εθνικό επίπεδο ε, ε, λόγω της απλούστευσης η οποία ενέχεται για μας ήταν δύσκολα τα πράγματα αλλά για τα κράτη-μέλη ελπίζω θα είναι πιο απλά. Όταν κ. Ολμπρέχτη και των υπόλοιπων συναδέλφων ήμουν κάπως απογοητευμένη γιατί αυτό που διαβάζω από την έκθεση είναι ότι να συνεχίσουμε όπως συνεχίσαμε για τα παλιά και για τα νέα πράγματα να υπάρξουν καινούργιοι πορεί. Είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα και παράλληλα κρίση επικουρικότητα για αυτά που αποτελεί, αυτά που αποτελούν αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέμα ευρωπαϊκά, θέματα ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τόσο μεγάλε φιλοδοξίες για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Το θέμα της ε, για τους νέους, κοιτάξουμε τα θέματα επικουρικότητα. θα πρέπει να σταματήσουμε να μπλέκουμε τις αρμόδιότητες που τελικά να καταλήγει να μην είναι κανεί υπεύθυνο για τέτοια θέματα. Η αιρεσιμότητα, μου λείπει. Δεν τη βλέπω πουθενά, γιατί είναι πολύ σημαντική για πιο πολλά χρήματα. Και αν πραγματικά... Κυρία Καρδία Θάβαλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτη φορά συζητούμε πραγματικά σε βάθος το θέμα αυτό Έχοντα μπροστά μα όλε τι νομοδοτήσει, Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον Επίτροπο, με ορισμένα από αυτά που είπε δεν συμφωνώ πλήρω. Ε, μίλησε πριν από μένα η κυρία Γκρέσλε και μπορώ να πω ότι διαφωνώ με πολλά από όσα είπε. Για παράδειγμα για την επανεθνικοποίηση ενό τμήματο τη ΚΑΠ. Θα ήταν στρατηγικό λάθο από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οικονομικό λάθο, μια και πολλέ μελέτε δείχνουν, αποδεικνύουν ότι η κοινή αγροτική πολιτική ήταν πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο φτηνή από τις αντίστοιχες εθνικές, από το άθροισμα των εθνικών πολιτικών. Οι γεωργοί, οι αγρότες έχουν κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πολιτική. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπαναχωρήσουμε. Δεύτερο, η αιρεσιμότητα. Συζητείται εδώ και πολλά χρόνια, ιδιαίτερα με την κρίση των προσφυγικό και με τη ε, διαφωνία ορισμένων κρατών με την υλοποίηση των υποχρεωσεών τους ξαναμπήκε στο τραπέζι. Διαφωνούμε. Όλα τα κρατημέλη θα πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Και αν όχι, θα πρέπει να τιμωρούνται. Αλλά δεν συμφωνώ να τιμωρούνται μέσω του Ταμείου Συνοχής. Γιατί γιατί τι το ιδιαίτερο έχουν τα ταμεία συνοχής για να τα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να τιμωρούμε κάποιο κράτο μέλο. Πολύ δε περισσότερο που οι πόροι του πηγαίνουν στις περιφέρειες και τους Δήμους που δεν είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε κεντρικό εθνικό επίπεδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να μπαίνουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου τα ταμεία συνοχής για ένα λάθος το οποίο κάνει η ε, κεντρική κυβέρνηση. Ας βρούμε ένα άλλο τρόπο, ας, υποβάλουμε, ας επιβάλλουμε πρόστιμα, ε, όπως συμβαίνει και με, πολλά, με άλλες παραβάσεις ε, κρατών μελών. Ο Επίτροπος εδώ και μήνες αναφέρει την άποψή του για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και με νούμερα ε, λέει ότι το, το Brexit θα το αντισταθμίσουμε κατά 50% με νέους πόρους, το άλλο 50% θα πρέπει να προκύψει από μειώσεις. Ε, και επίσης λέει και κάτι άλλο, ότι θα μειώσουμε ε, τον προπολογισμό κάποιων προγραμμάτων χωρίς να επηρεάσουμε την απόδοσή τους. Αυτό εγώ δεν το βλέπω να μπορεί να συμβαίνει. Αν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν το είχαμε κάνει πιο πριν. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί δεν έγινε πιο πριν. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Το ερώτημα είναι τι θέλουμε, ποια προγράμματα θέλουμε να προασπίσουμε στο μέλλον. Σε ορισμένους τομείς ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει περισσότερα και το ε, συμβούλιο ε, το έχει προβλέψει και υπάρχουν και προγράμματα στα οποία οι πολίτες μας ζητούν να ε, αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Ας μην γελιόμαστε. Ευχαριστώ. Κυρία Βάιντερε, άκουσα τον κύριο Ότιγκερ και νομίζω ότι η Κομισιόν είναι στη σωστή άγουσα. Συμφωνώ και με τις προ, ε, της προτεραιότητας Ένωσης για την οποία μίλησε η κ. Σβάρμα, θέλω να προσθέσω το εξή. Η εσωτερική αγορά λειτουργεί καλύτερα. Ό,τι εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε ήδη κάνει πολλά, αλλά μπορούν να γίνουν πολλά και στο μέλλον. Έτσι ώστε η Ανατολική Ευρώπη να προσθέμενη αξία. Επίσης χρειαζόμαστε επενδύσεις στις ε, υποδομές με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, ε, το συνδρομικό δίκτυο το οποίο θα συνδέει τις χώρες Βαλτικής με, το, με την κεντρική και την νότια Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό επίσης. Οι ανάγκες είναι πολύ λογικό είναι πολύ λογικό ε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας υπέρ της ε, αμυντικής ένωσης. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τους συνάδελφους που ζητούν να υπάρξει μια πιο ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική και ισχυρή πολιτική συνοχής. Προφανώς και πρέπει να μιλήσουμε για την αναδιοργάνωση, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την απλούστευση των πολιτικών αυτών αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μείωση των πολιτικών αυτών γιατί θα ήταν ένα εξαιρετικό κακό μήνυμα για τους πολίτες. Για τη συνοχή θα ήθελα να πω ότι οι πολιτικές αυτές έχουν σχέση και με τις κλιματολογικές αλλαγές και με την ψηφιοποίηση η πολιτική της συνοχής είναι επίσης πολιτική αλληλεγγύης. Υπάρχουν θέματα στον προϋπολογισμό, το ένα είναι οι νέες προτεραιότητες και την άλλη η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι δυνατόν να βρεθούν εύκολες λύσεις για τα θέματα αυτά στο μέλλον. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος Λαμασούρ. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Έτιγκερ, αλλά ίσως οι συνάδελφοι Όλμπριχτ ε, και άλλοι να μπορούν να δώσουν μία απάντηση. Ο κύριος Έτιγκερ μας είπε ουσιαστικά ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας δεύτερος προϋπολογισμός στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μια συγκεκριμένη δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη, δυνατότητα για την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν τα ειδικά προγράμματα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, των διαφορετικών αλλαγών και της σύγκλησης ή μήπως όλα αυτά θα τα επιδιώξουμε στο εσωτερικό της πολιτικής συνοχής ε, στους εισηγητές. Θα μου επιτρέψετε παρακαλώ να πάρω το λόγο σε προσωπικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ για την και ενδιαφέρον γιατί μου εμπιστεύθηκατε την Προεδρία σας. Αλλά βλέπω ότι όταν δημιουργούνται κρίσεις, όταν δημιουργούνται απρόβλεπτες καταβαρύνουν δημοσιονομικά τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Αν υπάρξουν νέοι ήδη πόροι, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε επίπεδα, δώσουν περισσότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας ελαφρύνουν όμως από την τυραννία της δίκαιης επιστροφής που θέτουν σε αντιπαράδοσουν περισσότερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας ελαφρύνουν όμως από την τυραννία της δίκαιης επιστροφής που θέτουν σε αντιπαρίσεις ε, η κοινή αγροτική πολιτική, συνοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι εκεί δεν θα πρέπει να δούμε και τα ποσά και ε, να κάνουμε ποιοτικέ επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν τους επόμενους μήνες το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε. Δεν λέω ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα εύκολο. Αμέσιο το οποίο μας αναιρεί κάθε δυνατότητα ευελιξίας. Τώρα για την προστιθέμενη αξία. Εγώ ε, πούμε ότι κινούμεθα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Κάποια τμήματα της κυριαρχίας μας δεν μπορεί να ασκηθούν πλέον σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο τρόπο σήμερα παρά μόνο εάν ασκηθούν σε ευρωπαϊκό. Οπότε μήπως θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη που μεταφέρουν λάσεις και εδώ ακριβώς ίσω να μπορέσουμε να αποδείξουμε τη ΦΠΑ, την συγγνώμη προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν πολύ παραγωγική. Ε, πράγματι ήταν λίγο έντονη, εντάξει δεν ε, χύθηκε αίμα, αλλά ήταν αρκετά έντονη η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Σάρβα, μα εδώ είμαστε κοινοβούλιο, δεν είμαστε συμβούλιο, δεν είμαστε επιτροπή, να χρηματοδοτηθούν και ε, εφόσον υπάρχουν θα πρέπει να τηρήσουμε τα υπεσχημένα σύμφωνα και με το 3.11 της συνθήκης. Να βάλουμε μια κόκκινη αλλά αυτό είναι η σωστή χρηστή διαχείριση. Πρέπει να είμαστε λογικοί. Δεν είναι λογικό να ανακοινώνουμε μια νέα ανάγκη καθημερινά και να μην προβλέπουμε τους πόρους που απαιτούνται για την κάλυψή της. Συνεπώς λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε στο μέλλον και για τα, τα συγκλίνη θα πρέπει να αυξηθούν τα μια μέρα στην άλλη. Εγώ προσπαθώ να είμαι λογική, προφανώς δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Αλλά νομίζω ότι οι ανάγκες σύγκλησης ε, εξακολουθούν να υπάρχουν, οπότε γιατί να τις μειώσουμε. Τώρα πάντα για λοιπόν τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πραγματικά παράλογο για την ΚΑΠ. Το ίδιο πράγμα. Αν πράγματι, βλέπω εδώ ότι οι συνάδελφοι που μίλησαν γι' αυτό φύγανε, ε, νομίζω ότι και για τους οικολογικούς μας στόχους μέσω της γεωργίας χρειαζόμαστε να μάθει γιατί δεν απαγορεύεται να επανεθνικοποιήσουμε τη γεωργία. Μα τότε σε αυτή την περίπτωση θα πέσουμε πάλι σε ένα σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ μας και θα οξύνουμε τον ανταγωνισμό και αυτό είναι εις βάρος συνολικά της οικονομίας μας. Είδα και μία επιστολή των γαλλικών αρχών στην Επιτροπή όπου λέγεται «Φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεπώς δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες δαπάνες, σώπα τώρα». Ε, πράγματι φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. τις ανάγκες, εφόσον τις διαπιστώσαμε υπάρχουν οι ανάγκες αυτές. Και για το θέμα της άμυνας τώρα, γιατί τέθηκε. Προφανώς και είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Προφανώς και να υπάρξει ένα κομμάτι διαχείριση, υπάρξουν νέοι πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία το μα μείνατε κάτω από πέντε λεπτά, δεν το είχα διευκρινίσει ότι καθένας από εσά έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά. Ο κύριος Όλμπριχτ έχει το λόγο. Καλό είναι να μας τα λέτε πριν και όχι μετά, λέει ο κύριος Όλμπριχτ. Για να μην είμαι και πολύ πολιτικά ορθό. αν να πω ότι το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, το συζητάμε, τι συζητάμε σήμερα, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τη δική μας πρόταση. Γιατί Σήμερα συζητάμε από πολλές ε, συναντήσεις και να πω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πραγματικό στην Επιτροπή. Τώρα λοιπόν η προτάση συζητάει τι θα κάνει για την προτάση της το Μάιο, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ε, φιλοδοξίες από τους επιτρόπους για το τι θα γίνει το Μάιο και παρακολουθούμε τα πράγματα με να κάνουμε μια πρόταση, να υποβάλουμε μια πρόταση επιτάπητος, η οποία θα είναι και φιλόδοξη, γιατί είμαστε κοινοβούλιο, και ρεαλιστική. Είμαστε κοινοβούλιο, λοιπόν. Είναι πολιτική αυτή η κίνηση. Τι λέμε λοιπόν, ότι τώρα είναι η σειρά σα προς το Συμβούλιο. Τι θέλετε να περικόψετε. Γιατί σύμφωνα με τις δικέ μας αναλύσεις, αν πει του Συμβουλίου να αποφανθεί και να μας πει ότι «Α, εντάξει, δεν συμφωνούμε». Ε, θέλουμε να σταματήσουμε αυτή την παράδοση του προτείνουμε ένα ποσοστό 1,5% αυτό προκύπτει από την ανάλυση. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να συζητήσουμε την πρόσθετη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί θα πρέπει να συζητήσουμε πιο πολύ το περιεχόμενο των πολιτικών. Αυτό που είπε και η κυρία Τόμα. Το θέμα του τι αποτελεί πραγματικά η γεωργική πολιτική. Τι είναι πραγματικά η γεωργική πολιτική. Είναι ένα τμήμα της οικονομίας. Είναι η παραγωγή είναι θέμα τη αλληλεγγύη, όχι τη οικονομία. Τώρα θα πρέπει να τα κοιτάξουμε τα ερωτήματα αυτά, αν θέλουμε κάτι να αλλάξει, γιατί κάτι πρέπει να αλλάξει. Το θέμα λοιπόν ε, του πώ θα αλλάξει είναι αυτό που είπε ο κ. Χόγκαν. Τι είναι συνοχή, ίσω έχει έρθει το πλέον του χρόνου να απαντήσουμε και αυτή την ερώτηση. Δεν υπάρχει γενικώ πολιτική συνοχή. Ο συγκεκριμένο χαρακτήρα ε, τη συνοχή δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο, αλλά με τη μέθοδο. Η μέθοδο είναι κοινή διαχείριση. Όταν λοιπόν επικρίνουμε τη δαπάνη των μέσων, επικρίνουμε το περιεχόμενο ή τη μέθοδο. Επικρίνουμε το πώς δαπάνονται τα χρήματα. Το θέμα είναι το τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Αυτό είναι θέμα περιεχομένου και συγχαίουμε τη μεθοδολογία με το περιεχόμενο. Χρειαζόμαστε τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στη συνοχή. Ναι, θέλουμε κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη γιατί όλο και πιο πολύ την περικόπτουμε με το ΣΕΦ ενισχύονται. Το κεφάλαιο χωρίς τη συνοχή αυτό θα αλλάξει παντελώς Εκβάτρων την πολιτική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν αν συζητάμε λιγότερη συνοχή εννοούμε λιγότερη συνοχή γιατί. Για τις υποδομές, για τις μεταφορές. Άρα θεωρώ ότι αυτό που λέμε σήμερα να μας το εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το αναφέραμε και με την κυρία Γκαρτά Σαμπάλα. Αυτό το 50%, 50% Πώ γίνεται και μετά να κάνουμε περικοπέ στην πολιτική συνοχή κατά 15%. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά. Πώ συνδυάζονται, πώ θα καταστεί δυνατό αυτό και πώ θα γινεται δηλαδή περιμένω σιγά σιγά και φτάνω τα πέντε λεπτά που μου δώσατε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν επικρίναμε την πρότασή μα στην παρούσα φάση. Την κρατική θα την αντιμετωπίσουμε τι ερχόμενε ημέρε. Τώρα είμαστε σε πρώτη φάση ακόμα, είμαστε αντιτεθειμένοι να συνεργαστούμε να ξεκινήσουμε μια σοβαρή συζήτηση, όχι μόνο για τα αριθμητικά στοιχεία, για το μέλλον συνεισφορές σας. Και οι δύο εκθέσεις κινούνται παράλληλα με το διάγραμμα και έχουν κοινό στόχο να ενθαρρύνουν τον Oettinger και την Επιτροπή στις προτάσεις που θα καταθέσουν το Μάιο. Για μένα το πιο συνερπαστικό σήμερα ήταν που άκουσα τους Γάλλους συναδέλφους να εκφράζουν ε, σκεπτικισμό για την κοινή αγροτική πολιτική. Ε, επανάσταση έκτασης Κοπέρνικου θα έλεγα. Το συμπεραίνουμε αυτό ελήψη του Επιτρόπου, αλλά οι ήδη πόροι ε, αποτελούν ένα θέμα ειδικότητα άλλωστε και του Ελλάδα Λαμασούρο, ο οποίος είναι παλέμαχος και θα συμφωνούσε ότι είναι πλέον, θα είναι πλέον πιο απλό να συζητήσουμε το θέμα των ιδιαίτερων πόρων χωρίς ε, τον ε, Κάμερον και χωρίς το θέμα της ε, λιτότητας που επαπειλούσε στο παρελθόν το 2012 και 2013. Αλλά και πάλι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σόφρονες, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική χρονιά και δεν μπορούμε ότι ένα ευρώ που πηγαίνει στις Βρυξέλλες είναι ένα ευρώ το οποίο ε, εξοικονομείται από τον εθνικό προπολογισμό, για παράδειγμα, στην αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση. Υπάρχουν λοιπόν δαπάνε χωρί να υπάρχουν και οικονομίε σε εθνικό επίπεδο. Ούτε μπορούμε να υποσχεθούμε τη μεσονομική αμοιβαιότητα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. εννοούμε την ε, ονομαστική αξία του προπολογισμού χωρί τη συμβολή των Βρετανών. Άρα θα πρέπει να είμαστε και κάπως πονηρή στο θέμα αυτό. Ο Έττιγκερ έχει στρομολογηθεί προς τα πλαστικά. Και για το ETS, το σύστημα εμπορία ρήπων. Για το σύστημα εμπορία ρήπων. Είναι τεράστια η τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μου προκαλεί έκπληξη δις ευρώ. Αυτό δεν είναι πολύ και θα μειωθεί και ως πόσο στο μέλλον, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ ε, φιλόδοξους στόχους για τη μείωση μα του και ε, πέρασε από βαριά διαπραγμάτευση. Καλύπτει και την Ορβηγία το ETS. Αν το επιλέξουμε αυτό, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε λούσα ήταν να αποφύγουμε το περιβαλλοντικό dumping και τον φόρο προσαρμογής των άνθρακα για να είναι ίση όρη ανταγωνισμού. Gérard euh, τελευταίος στη λίστα. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη συζήτηση, έκαναν σχόλια και κριτική. Καταρχήν είμαι ουδέτερος σε ό,τι αφορά τους ηγητές του πολιτισμού νομικού πλαισίου, έτσι κι αλλιώ και οι ίδιοι ήταν ουδέτεροι σε ό,τι αφορά τη δική μα έκθεση. Οπότε το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Δύο λόγια μόνο. Συμφωνώ με την φιλοδοξία του. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθορίζει τη σχέση ανάμεσα στι πιο ανεπτυγμένε χώρε και τι λιγότερο. Να πω όμω το εξή. Νομίζω ότι είναι θεμητό να αναρωτηθούμε για το τι τοποθετούμε εντός της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο. Μόνο έτσι θα δούμε ποια είναι τα ποσά τα οποία χρειάζονται για την πολιτική συνοχή. Δεύτερον, σχολιάζοντας αυτό που είπε ο Γιάννους για την φορολογική ουδετερότητα. Πρέπει, ε, συγγνώμη, τη δημοσιονομική ουδετερότητα, πρέπει να την κατοχυρώσουμε. Γιατί αν αύριο χρειαστεί να αυξήσουμε τους πόρους και κάθε φορά που αυξάνονται οι ήδη πόροι πρέπει να μειώνονται οι εθνικές φορές, δεν θα έχουμε πρόσθετους πόρους. Αν κάθε φορά γίνεται μία αντιστάθμιση, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μειωθούν οι εθνικέ φορέ κάθε φορά που εισάγουμε ένα καινούριο ίδιο πόρο, αλλά όχι κατά αντίστοιχο ποσό. Όχι κατά το ίδιο ποσό. Τώρα, το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών, εμπορία εκπομπών, ε, είναι πιστεύω ένα από τα πιο σημαντικά και πιο δύσκολα καθόδη προβλήματα. Πρέπει να μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Γιατί πολλές πολιτικές ομάδες θέλουν συνένεση, θέλουν να εγκριθεί, αλλά θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπο. Στο κύριο Σαβραμά. Να πω το εξή. Συμφωνώ μαζί του που λέει πως, πως πρέπει να έχουμε την γενναιότητα να πούμε εφόσον έχουμε κάποιες προτεραιότητες πρέπει να έχουμε και τα αντίστοιχα μέσα. Και σε ένα, κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αποφασίσουν ότι αξίζει τον κόπο. Πρέπει να πάμε να τους πούμε ξεκάθαρα αυτά χρειαζόμαστε αφού αυτά θέλουμε να κάνουμε. Να πω όμως το εξή. Αν το πούμε αυτό, αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να μας δώσουν τίποτα. Να το πούνε οι, οι, οι, οι υπέρμαχοι της όμως πονδιοποίηση της Ευρώπης, ναι. Αλλά αν θέλουμε να βάλουμε τους ίδιους πόρους στην διαπραγμάτευση του, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο αν έχουμε ισχυρή πλειοψηφία. Γιατί αλλιώς θα σπάσουμε τα μούτρα μας στο Συμβούλιο. Οπότε, η πρώτη μου προτεραιότητα, και μπορώ να κάνω υποχωρήσει για αυτό το θέμα, είναι να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις μας. Αν θέλετε να γίνουν κάποιες προσαρμογές, διορθώσεις κλπ. υποβάλλετε προτάσεις, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε την πιο ευρία, δυνατή συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας περάσω. Πρόεδρος, δεν θέλω να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση βέβαια, αλλά να, σχολιάσω αυτό που είπε ο κ. Ντεπρέ. Πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί ο προπολογισμό χωρί να αυξηθεί η φορολόγηση. Μειώνοντα όσο αυξάνουμε. Ναι, λέει ο κ. Ντεπρέ. Χτες το βράδυ έγινε μια συζήτηση στο πλαίσιο της ε, δέκατης ετήσιας ε, συνόδου για την Ευρώπη το διάστημα. Ε, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι υπερεθνικό είναι το διάστημα. Υπάρχουν όμως κάποια ποσά τα οποία επενδύονται σε εθνικό επίπεδο και 14-15 δισεκατομμύρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ας με διορθώσει η Μόνικα αν κάνω λάθος, ήταν παρούσα. Αν θέλει κανείς να είναι πιο αποτελεσματικός στον τομέα του διαστήματος, με πρωτοβουλίες που επηρεάζουν όλους τους Ευρωπαίους, Κοπέρνικος, Γαλιλαίος κλπ, θα πρέπει να είμαστε να πάρουμε μία απόφαση. Ε, χρειάζεται να θέσουμε σε κοινή χρήση τους εθνικούς προπολογισμού που επενδύονται σε αυτό το κλάδο, τον τομέα. Ή αρκεί η κατάσταση έτσι οτι οπως είναι. Δηλαδή τα κράτη να βάζουν στον, στον, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό μόνο ότι περισσεύει από τους εθνικούς τους. Αυτό θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες. Ο προπολογισμό αυτή τη στιγμή είναι ακατανόητος. Το 80% στην πράξη αναδιανέμεται στα κράτη-μέλη. Τι μένει, μένει ένα 20% για τα, τις υπερεθνικές δράσεις. Αυτό πραγματικά είναι ευρωπαϊκό. Μόνο η τελωνιακή δασμή είναι ο πραγματικός πόρος μας και τι κάνουμε στις ε, συμφωνίες ελεύθερων ανταλλαγών που υπογράφουμε τη μία μετά την άλλη ε, καταργούμε τους τελωνιακούς δασμούς. Απ' την άλλη μεριά στην κοινή αγροτική πολιτική δίνουμε ε, επιδοτήσεις στους ε, κτηνοτρόφους μας και από την άλλη μεριά τους θέτουμε σε κατάσταση πτώχευσης υπογράφοντας συμφωνίες ελεύθερων ανταλλαγών, ε, ελεύθερων συναλλαγών με την Νότιο Αμερική. Ε, του χρόνου έχουμε εκλογές. Και ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι έτοιμος πριν γίνουν οι εκλογές. Ε, με ορισμένοι από εσά συμμετείχατε στη διαπραγματεύση του 2013 και τι έγινε. Ε, είναι, συνέβη κάτι πρωτοφανέ. Ε, πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό. Ενδιαφέρουσα θα είναι η επόμενη περίοδος. Αυτά σε ό,τι αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τις, ε, το σύστημα ιδιών πόρων. Κύριε Τωμά, μια ερώτηση, Πρόεδρε, για την ημερήσια διάταξη. Ε, για αυτές τις δύο εκθέσεις. Οι τροπολογίες θα υποβληθούν προθεσμία υποβολής τροπολογιών 31 Ιανουαρίου. Και Ψήφο στην Επιτροπή Προπολογισμών στη συνάντηση 20, της 21ης και 22ης Φεβρουαρίου, έτσι ώστε στην Ολομέλεια να γίνει συζήτηση και ψηφοφορία τον Μάρτιο στο Στρασβούργο. Ο λόγος τώρα στον Ντανιέλε Βιώτη, Γενικό Εισηγητή για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες προπολογισμού του 2019. το συζητήσαμε ε, εκτεταμένα. Μάλλον έχουμε συζητήσει θέματα τα οποία δεν απέχουν και πάρα πολύ από τα θέματα αυτά που άπτονται τη έκθεσή μου. Δεν χρειάζεται να επισέλθω σε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά το κείμενο, γιατί οι συνάδελφοι τι επόμενε ημέρε ε, θα έχουν την ευκαιρία να το διαβάσουν και ενδεχομένω ε, να ασκήσουν κριτική μέσω τροπολογιών. Αλλά να εκφράσω κάποιε σκέψει γενικότερες σε ό,τι αφορά και τις παιδικές προοπτικές. Θα ήθελα να το βασικά, οι οποίες, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τον προπολογισμό, εξωγενή στοιχεία. Το ε, πρώτο κομμάτι είναι φυσικά η συζήτηση για μας πλησιάζει όλο και περισσότερο το φάντασμα του Brexit ο προϋπολογισμός λοιπόν για το 2019 θα χαρακτηρίζεται που είναι η άλλη αρμόδια αρχή για τον προϋπολογισμό. Εμείς ε, βλέπουμε ποιες είναι οι προσδοκίες των πολιτών λαϊκισμό. Δεν είναι αυτός σκοπός αυτή η προσπάθεια. Αλλά θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη ενωμένη, μια Ευρώπη η οποία έχει διασφαλίσει 70 χρόνια πολιτικές. Ε, μιας και πιστεύω ότι υπάρχουν τμήματα του συνόλου των πολιτών οι οποίοι έχουν χτυπηθεί περισσότερα πίσω εδώ και τον συνάδελφο μου Ρεσάν για αυτά τα οποία έκανε πέρυσι. Ράιζον και τα λοιπά. Κάναμε μια καλή δουλειά. Νομίζω ότι από τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ακόμα περισσότερο σε θέματα, σε πιο θαραλέη, σε τέτοιου είδους θέματα στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τους Νέους, ε, στη στήλη της οικονομίας μας. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη, νομίζω, να εργαστούμε ακόμα περισσότερο για το κοινωνικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο θα έλεγα φάνηκε στις συζητήσεις οι οποίες κάναμε σήμερα το πρωί για τον προϋπολογισμό. Πριν λίγες μέρες ή χθες ίσως ο πρόεδρος Πρόντι είχε παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις λεγόμενες κοινωνικές υποδομές στα πλαίσια της, των ψηφιακών οικοδομών, των ε, υποδομών γενικότερα, υπάρχουν και οι κοινωνικές υποδομές. Και θα πρέπει να είμαστε ικανοί, μιας και εμείς είμαστε η συνδετήρια δύναμη ανάμεσα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ευρωπαίους πολίτες και μέσα στη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό θα μπορέσουμε νομίζω να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ε, ε, γίνει πραγματικότητα αυτό το ε, σχέδιο ενίσχυσης του κοινωνικού τομέα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο άπτεται όλων των προηγούμενων βέβαια, δύο στοιχεία μάλλον περισσότερο και μετά θα προσπαθήσω να κλείσω για τη μετανάστευση Νομίζω ότι υπόθηκε και από τους προηγούμενους. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην μετανάστευση, την άμυνα και την ασφάλεια. Το θέμα της μετανάστευσης θα πρέπει να το δούμε σαν ένα υποεξέλιξη, υποανάπτυξη πρόβλημα και θα υπάρξει μάλιστα υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ε, δεν συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Έτιγκερ στην ε, παρουσίασή του σήμερα το πρωί είπε ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, προστατεύσουμε τα θαλάσσια μας σύνορα. Σας ομολογώ πρόεδρε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Πάρα πολύ περίπλοκο όχι μόνο γιατί είναι τεχνικά περίπλοκο, αλλά γιατί θα πρέπει και σε επίπεδο ανθρωπιστικό να, να υπερασπιστούμε τα σύνορα αυτά. Εμείς σαν Ευρώπη δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα χωρίς την αλληλεγγύη, χωρίς τη φροντίδα προς τον άλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, σε σχέση με όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε ιδιαίτερα στην πρόβλεψη των οικονομικών πόρων. Πέρυσι έγιναν κάποια πρώτα μικρά βήματα, ανοίγοντας μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Εάν πράγματι εμείς είμαστε ικανοί να επενδύσουμε εκεί όπου γεννιούνται τα προβλήματα της μετανάστευσης, εκεί που γεννιέται η φτώχεια, τότε ε, θα μπορέσουμε νομίζω σε χρόνο εύθετο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να βοηθήσουμε να μειωθεί το μέγεθός του. Τώρα, σε επίπεδο μεθοδολογικό, θα ξεκινήσω ε, όμως με ένα κομμάτι που άπτεται του περιεχομένου. Όπως συνέβη και πέρυσι και όπως συζητήθηκε και σήμερα το πρωί σε σχέση με το επόμενο πολιετές, νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα πάνω στο οποίο θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ενότητα μεταξύ μας σαν κοινοβούλιο, είναι ότι οποιαδήποτε νέα ιδέα ε, εκπέμπει το Συμβούλιο και οποιαδήποτε επιθυμία και αν έχει το Συμβούλιο για νέες πολιτικές, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συνδέονται με νέου τύπου επενδύσεις. Και σε σχέση με το Συμβούλιο των θέσεών μας και τη συμφωνία την τελευταία στιγμή, αλλά να κάνουμε μια πραγματική προσπάθεια διαβούλευσης, ε, συνδιαμορφώνεται ε, το ημερολόγιο και το χρονοδιάγραμμα της ε, συνδιαλλαγής. Είναι σαν το Πάσχα, κανένας ποτέ δεν καταλαβαίνει πότε θα είναι. Τελειώνω λέγοντας ότι αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνω. Η πρόθεσή μου είναι να α, ταυτόχρονα και εγώ θα προσπαθήσω να επιδιώξω να κάνω το ίδιο μετά τον μήνα Μάνιο, Μάιο όταν θα έχω το κύριε Γιώτη. Ευχαριστώ και για τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες μας προτείνετε. Έδωσε τέσσερις συνδιαλλαγές. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει μία θεατρικού τύπου διάσταση για δύο εβδομάδες, σαν παράδειγμα, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πηγαίνει στη συνδιαλλαγή μερικές φορές ε, χωρίς να εκτά ουσιαστικά. Εσείς είπατε ότι θα προσπαθήσετε να το αποφύγετε φέτος. Θα προσπαθήσουμε και εμείς μαζί σας να βελτιώσουμε τη μέθοδο έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η συνδιαλλαγή αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι θέλει και να μειώσει το ε, Χολμάιερ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και για τις νέες ε, κατευθυντήριες γραμμές και για το κείμενο. Πρόκειται για θέματα για τα οποία έχουμε αγωνιστεί από κοινού με πολύ πάθος και με μακρό χρονικό διάστημα. Οι συζητήσει για το Erasmus Plus, οι συζητήσει που έκαναμε με τα κράτη-μέλη για το αποτέλεσμα, μεγάλο αντίκτυπο για τους νέους. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω για την ε, πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Νεολαία. Διάβασα και εγώ την έκθεση του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συνεδρίου θα ήθελα να ξέρω. Αυτό φυσικά για το 2019 προσπαθήσαμε σε κάθε περίπτωση, κάθε χρονιά να προχωρήσουμε όσο μπορούσαμε, όσο μας θα το επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά φροντίζουν καλύτερα και τους νέους και όλους τους εργαζόμενους να έχουμε πιο πολλές θέσεις απασχόλησης και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εστία. Θέλουμε να διαμορφώσουμε τις υπηρεσίες μας με αναλογικό τρόπο, γιατί σε διάφορες περιπτώσεις βλέπουμε διάφορες υπηρεσίες, είτε είναι αυτές που αναπτύσσονται με γουργού, έχουν δυσπιστία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα φορολογικά μέτρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι πολίτες βασικά δυσπιστούν απέναντι τώρα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Τηρούσαμε πάντα και τα ε, την επικουρικότητα και τις συνθήκες της Λισαβόνας. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα συστήματα υφιοποίηση επίση, και χθε στην διάσκεψη το ακούσαμε αυτό, δεν είναι γενικά κάτι αρνητικό. Η ψηφιοποίηση θα σημαίνει και πολλέ καινούριε θέσει απασχόληση, αλλά θα έχει και αρνητικό αντίκβαληση, αλλά και την πρόσβαση του κόσμου στο δικτύο, προκειμένου ο κόσμο να έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την ψηφιοποίηση, για να την αξιοποιεί όταν μιλά για την πρόσβαση στην ώρα εργασία για τι γυναίκε. Νομίζω κοιτώντα και τον προπολογισμό του δύο σημαντικό. Η επικορικότητα σύμφωνα με την συνθήκη της Γενέβης θα πρέπει να είναι και απέναντι στα θετικά μέτρα, γιατί σωστά λέτε ότι θα σταματήσουν τα θετικά μέτρα και στη συνέχεια όλοι οι θέματα άμυνα, προφανώ η ομάδα μα έχει κάποιε αμφιβολίε. Ε, νομίζουμε ότι αρκετά ασφαλή είναι πια ο κόσμο. Σα προσπέρασα γιατί έφευγε ο συνάδελφο. Δεν ήξερα ότι είναι δική μου σειρά, λέει ο κ. Δεπρέ. Εν πάση περιπτώσει, μου αρέσει η έκθεση βιώτη. Πρώτον, διότι είναι σύντομη. Σε σχέση με άλλες εκθέσεις που δείχνουν να είναι ατελείωτες. Είναι καλά δομημένη, σαφής, ε, εντάξει, ευανάγνωστη, έχει σχετικά σαφείς προτεραιότητες, πολύ σαφείς προτεραιότητες θα έλεγα. Ενδεχομένως λίγο υπερβολικά σαφείς μερικές φορές λέει πρέπει ο προβλημό 19 να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. κατά κύριο λόγο. Τώρα το κατά κύριο λόγο, primarily, είναι ίσως λίγο υπερβολική έκφραση, εν πάση περιπτώσει. Καλό το μήνυμα, το πολιτικό μήνυμα που βγαίνει. Για την προτεραιότητα και να θέσουμε και άλλους στόχους, όπως για παράδειγμα να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα των νέων, τα προσόντα τους, να, ικανοποιηθούν όλοι οι επιλέξιμοι, όλες οι επιλέξιμες ε, αιτήσει. Η αρχή κρατών στη διαφορά ανάμεσα στο, στις αιτήσει και σε αυτούς που μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον προπολογισμό, καταλαβαίνω πόσο μεγάλη, κατάλαβα πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση. Τώρα, για την